Good afternoon, colleagues, and uh, Καλησπέρα, συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε ξανά στην Επιτροπή μας ε, και καλή χρονιά. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, ε, η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. Για τα γλωσσικά δεν έχουμε σήμερα κροατικά, δανειζικά και ιρλανδικά. Έχουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 5ης Οκτωβρίου. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνονται. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 4, αποστολή στην Τίνιδα, στην Τινησία, τον Σεπτέμβριο 18 21 και έχουμε κάποιους συναδέλφους εδώ από την, Ισία μεταξύ των οποίων και ο πρέσβης η αντιπροσωπεία μας αυτή ήταν πολύ σημαντική στόχο είχε να κατανοήσουμε καλύτερα όχι μόνο την συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τινησίας αλλά και την σχέση μας με την Λιβύη όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων και την διαχείριση της μετανάστευσης και έτσι συναντηθήκαμε με ενδιαφέρομενα μέρη και στις δύο χώρες, ε, υφυπουργό εξωτερικών, εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, εκπροσώπους και των δύο χωρών και των διαφόρων υπηρεσιών του ΟΗΕ, την Ιταλική και Λιβική Ακτοφυλακή, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η σημερινή μας συζήτηση λοιπόν λαμβάνει χώρα με βάση το σχέδιο έκθεσης στο οποίο καλούνται να συνεισφέρουν όλοι οι συνάδελφοι, γραπτός ή αν θέλουν και σήμερα. Ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τις αρχές της χώρας και τον τον πρέσβη για την υποδοχή της αντιπροσωπείας μας, πολύ σημαντικής αντιπροσωπείας, ειδικά για να καταλάβουμε τις σχέσεις την νησία και Λιβύης. Είχαμε πολύ καλή πρόσβαση στα άτομα τα οποία επηρεάζονται βεβαίως από την κατάσταση αυτή. Θα ήθελα τώρα να πούνε οι συνάδελφοι που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία δύο λόγια, αν θέλουν. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάρει τον λόγο. Αν δεν θέλει κανείς, Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Μαρή Κριστίν Βερζιά τότε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά που λέμε στην έκθεση της αντιπροσωπείας μας. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια σημεία που κατά τη γνώμη μας ήταν σημαντικά. Καταρχήν, η αντιπροσωπεία μας πρώτα απ' όλα ασχολήθηκε με την κατάσταση στη Λιβύη, γιατί αρχικά έπρεπε να πάμε στη Λιβύη. Κάτι τέτοιο κατέστη αδύνατο για λόγου ασφαλείας. Οπότε οι φόβοι που είχαμε για την κατάσταση στη Λιβύη δυστυχώς μάλλον επιβεβαιώθηκαν. Δηλαδή η πραγματικότητα της κατάστασης των μεταναστών κυρίως, αλλά και της κατάστασης ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικά σε αυτή τη ρηβαγμένη χώρα ε, μας θορύβησαν ιδιαίτερος και επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες μας και μάλιστα από την ε, ονομαζόμενη επίσημη κυβέρνηση της Λιβύης είχαμε και την επιβεβαίωση ότι ελέγχει μόνο ένα ελάχιστο τμήμα της επικράτειας της χώρας αυτής. Και παρόλο που η Λιβική ε, το φυλακή έστειλε κάποιους εκπροσώπους της στην την είδα στην Τινησία, στη που είχαμε, μας ενημέρωσε ότι ακόμη και η Λιβική Ακτοφυλακή ελέγχει μόνο ένα ελάχιστο τμήμα των Λιβικών ακτών. Και μάλιστα έκτοτε η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Και έχουμε αλλεπάλληλες εκθέσεις και αναφορές για την επιδείνωση της κατάστασης, παρόλο που οι κυβερνήσεις μας έλαβαν κάποια μέτρα που είναι μονόπλευρα, δηλαδή στέλνουν προς την ήγυρα κόσμο με κίνδυνο να αποσταθεροποιήσουν το βόρειο Ήγυρα χωρίς να αναλαμβάνονται κάποια μέτρα ώστε σημαντικό του πληθυσμού που βρίσκεται σε λιβικό έδαφος να έρχεται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επικράτηση, σε ευρωπαϊκό έδαφος, ευρω... έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, συνεχίζουμε τις επαναπροωθήσεις ε, ε, των σκαφών προς τη Λιβύη και ε, έχουμε και ένα κέντρο κλήσεων στη Λιβύη με στόχο να αποσυφορήσει το Ιταλικό κέντρο κλήσεων αλλά αυτό έχει μείνει ακόμη στα χαρτιά ακόμη αυτή η πρόταση. Δεν έχει υλοποιηθεί. Κάτι που μας ανησυχεί. Γιατί αν δεν έχουμε ε, κλήσεις ε, από τη Λιβύη καθόλου. Και παραμένει η Λιβύη μία ζώνη όπου δεν επικρατεί ο νόμος και το δίκαιο. Επίσης, πολλά ακούσαμε για τα μέτρα που θα ληφθούν εις βάρος αυτών που παραβιάζουν τα δικαιώματα των μεταναστών στη Λιβύη. Και εκπρόσωποι των διεθνών οργανώσεων που συναντήσαμε μας είπαν ότι δεν υπάρχει ε, δικαστικό σύστημα, απονομή δικαιοσύνη στη Λιβύη και δεν υπάρχει δυνατότητα ε, υποβολής μήνυσης ή άσκηση προσφυγής εις βάρος ε, όσων διαπράττουν αδικοπραξία εις βάρος των μεταναστών για μας είναι θεμελιώδεις αρχές ε, του δικαίου, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να, να ισχύσουν. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ της στιγμής πραγματικότητας που επικρατεί στη Λιβύη και των α, ε, ε, ωραίων λόγων που ακούμε μερικές φορές μέχρι και το Δεκέμβριο εδώ. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ θεωρίας και πραγματικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να εγκύπτουμε στο θέμα αυτό με αμύωτο ενδιαφέρον. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Τινησία, γιατί στην Τινησία πήγαμε και φυσικά κάναμε έναν απολογισμό και της κατάστασης των μεταναστών στην Τινησία και ε, το κύριο στοιχείο είναι ότι ε, εξαιτίας και της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής η Τινησία γίνεται από χώρα απόδημων μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής μεταναστών Φέρουμε λοιπόν και εμείς την ευθύνη να βοηθήσουμε την, Τινησία να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Επίσης στην Ισία έχουμε κάποιες μαύρες λίστες για νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα που μπορεί να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ισία στην δίνη κατάσταση που αντιμετωπίζει και διανύει σήμερα. Δύο είναι τα στοιχεία από την κατάσταση στην Τινησία που με εντυπωσίασαν το πρώτο είναι η ανάγκη η χώρα αυτή, την Ισία, να προσαρμόσει το νομοθετικό της μηχανισμό και μάλιστα έχουν ήδη κατατεθεί πολλά νομοσχέδια στο γραφείο της ε, την Ισιακής Βουλής και μάλιστα με τους ομολόγους μας ε, συζητήσαμε αυτή την ε, ανάγκη επιτάχυση της προσπάθειας ώστε να υιοθετηθούν σχετικές νομοθετικές πράξεις και να έχουν κάποια δικαιώματα όσοι, αφικνύονται, όσοι μετανάστες αφικνύονται στη Δινησία. Συναντήσαμε και εκπροσώπους μεταναστών που μας είπαν ότι είναι πολύ λεπτή η θέση τους, γιατί έχουν ε, καταδικαστεί σε βαρύτατα πρόστιμα λόγω της ε, παράτυπης παραμονής τους σε την Ισιακό έδαφος και μερικές φορές ε, εμποδίζονται και στην επιστροφή στην πατρίδα τους αν δεν καταβάλουν αυτά τα υπέρογκα πρόστιμα. Οπότε υπάρχει μια μικρή αντίφαση μεταξύ πραγματικότητας και πράξης ή θεωρίας. Θα πρέπει η Τινησία λοιπόν να αναθεωρήσει τη σχετική της νομοθεσία. Και σε ό,τι αφορά τους Τινήσιους που θέλουν να αποδημήσουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα πρέπει να στηρίξουμε ε, τη συμφωνία κινητικότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ισίας. Και αν είναι σωστές οι πηγές μου, ε, οι διαπραγματεύσεις έχουν αποτελματωθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απέρριψε η συμφωνία αυτή κινητικότητας να γίνει στο γενικό πλαίσιο της συμφωνίας με τις χώρες Μαγκρέπ Και μία συμφωνία κινητικότητας έχει δύο σκέλη. Το ένα σκέλος αφορά τις συμφωνίες επανειστοχής, με το οποίο δεν συμφωνώ, αλλά είναι ουσιαστικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει και ένα σκέλος που αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο ανοιχτό όσο θα, περιμένανε θα περίμεναν οι Και επίσης χρειάζεται και ένα σκέλος για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων, των τίτλων σπουδών, αυτό είναι σημαντικό διακύβευμα για τις χώρες του Μαγκρέπ γενικώ, αλλά και ειδικώ για την, Τινησία. Αυτά κύριε Πρόεδρε, εν γέννη για τα σημεία που κατά τη γνώμη μου ήταν σημαντικά στα πλαίσια της αποστολής Επιτροπής μας στην Τινησία. Ευχαριστώ. Thank you, Mary It's very comprehensive. Ευχαριστώ πολύ περιεκτικά αυτά που μας είπατε. Ο κύριος Τέτινα, που επίσης ήταν μέλος της ε, αντιπροσωπείας αυτής ε, και ανήκει στο ΕΛΚ. Σας ευχαριστώ. Κυρίε και κύριοι, εγώ θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, γι' αυτό παρακαλώ φορέστε τα ακουστικά σας. Εξοχότατε, ε, αγαπητοί προσκεκλημένοι από την Τινησία. Χαίρομαι ιδιαίτερως για την παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που έχουμε την ευκαιρία να συζητάμε για αυτή την ε, φοβερή κατάσταση, τη συγκλονιστική κατάσταση των μεταναστών και τη μεταναστευτική κρίση που αφορά και εσάς στην Τινησία και εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή όλων σε κάτι που με προβλημάτισε και με θορύβησε κατά τη διάρκεια της ε, αποστολής μας, της επίσκεψής μας στην Τινησία. Φυσικά συζητήσαμε και το θέμα της θυνησίας μεμονωμένα, αλλά μερικές φορές ε, ε, ε και τι συμβαίνει στη Λιβύη πέραν των συνόρων. Και το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις δύο χώρες. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε μία συνάντηση που είχαμε με ένα δημοσιογράφο Μάλιστα, ο συντονιστής ε, πρότεινε αυτή τη συνάντηση με τον Μάρκ Μίκαλεφ, αν δεν κάνω λάθος, ε, έτσι λέγεται. Ενδιαφέρουσα συνάντηση πρόκειται για έναν άνθρωπο που εργάστηκε στη Λιβύη ένα ή δύο χρόνια και κάλυψε κυρίως το θέμα της ε, διακίνησης ανθρώπων και το λέω αυτό γιατί στη Λιβύη υπάρχουν ε, δεκάδες ε, δημοσιογράφων που διαβιούν και εργάζονται εκεί, που παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να μας ενημερώνουν για την κατάσταση στη Λιβύη. Και ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πρεσβεία στην Τρίπολη. Έχει πρεσβεία στην Τίνιδα, αλλά όχι και στην Τρίπολη. Και ίσως ε, οι αξιωματούχοι από την Τινίδα θα μπορούν, ε, μπορούν και παίρνουν κάποια πτήση και πηγαίνουν για λίγες ώρες στην Τρίπολη, αλλά επιστρέφουν. Δεν παραμένουν αρκετά. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αντιμετωπίσουν αυτό το περίπλοκο πρόβλημα ως διπλωμάτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν επιδεικνύουν ούτε το ελάχιστο κουράγιο αντίστοιχο με αυτό που δείχνουν οι δημοσιογράφοι, όπως ο κύριος Μουκάλεφ, που διακινδυνεύουν τη ζωή τους με την παραμονή τους για μεγάλα διαστήματα στη Λιβύη. μπορεί να ακούγομαι απεσιόδοξο. Θα σα αναφέρω και μια άλλη συνάντηση που είχαμε, την συνάντηση με τον συνταγματάρχη Μασούντ, που είναι επικεφαλής του προγράμματος Διεθνούς Συνεργασίας για τη δημιουργία της Λιβικής Ακτοφυλακής. Κατά τη γνώμη μου, η συνάντηση αυτή ήταν ο φάρος που μας καθοδήγησε προς ε, τις επικοδομητικές συζητήσεις που θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και διαπραγματεύσει στη Λιβύη. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε θαραλέοι και να έχουμε κουράγιο για να ξεκινήσουμε αυτές τις συνομιλίες. Και μάλιστα η ομιλία του Σταματάρχη Μασούντ μας έδειξε ότι υπάρχει μια λύση στη συνεργασία. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κονδύλια εκπαιδεύει ε, στρατιώτες και μάλιστα ένας πολύ γοητευτικός ε, ακτοφύλακας από τη Λιβική Ακτοφυλακή μας διαβεβαίωσε ότι υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας χωρίς όμως το κουράγιο που θα πρέπει και το θάρρος που θα πρέπει να δείξουμε και σε προσωπικό επίπεδο μερικέ φορές για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα θα έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μα. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον άλλον να ζητάει τον λόγο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις αρχές της ε, Τινησίας. Γνωρίζω πως ε, είχαμε διάφορα μέλη, διάφορους βουλευτές ε, και όλοι όσοι πήγαν εκεί και εγώ μεταξύ αυτών εντυπωσιαστήκαμε και από την πρόσβαση που είχαμε και σε οργανώσεις και στους μετανάστες στην Τινησία. Ήταν μια συνήθιστη αποστολή γιατί αξιολογήσαμε αφενός την θέση της Τινησίας αλλά είχαμε και πρόσβαση στην Λιβύη, ένας ασυνήθιστος δηλαδή συνδυασμός, ε, κάτι το οποίο βεβαίως μας επέτρεψε να έχουμε μια συνολικότερη εικόνα και η Μαρή Κριστίνα έδωσε μια συνολική εικόνα θα έλεγα όλων των πτυχών. Η έκθεση νομίζω θα τα αναφέρει αυτά, αλλά νομίζω ότι επηρεάστηκε έτσι πολύ το έργο μας. Ευχαριστώ λοιπόν και τους δύο συναδέλφους ε, που μίλησαν ε, και ήταν στην αντιπροσωπεία. Για το άλλο θέμα τώρα, εάν δεν θέλει κανείς, ε, εάν δεν θέλει κανείς να μιλήσει από την αντιπροσωπεία της Τινησίας, ο κύριος Πρέσβης. Μία στιγμή. Ναι, ναι, όχι, παρακαλώ, μιλήστε τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα δευτερόλεπτα μόνο. Είναι προνόμιό μου και τιμή μου να είμαι εδώ Είμαι συνηθισμένος να έρχομαι σε συνεδριάσεις της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Το θεωρώ όμως κάθε φορά προνόμιο. Και μαζί μου έχω δύο υφυπουργούς. Τον Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και τον Υφυπουργό του Διεθνούς Εμπορίου. Και έχουν έρθει εδώ στα πλαίσια της ενίσχυσης των σχέσεων ε, Ισίας. Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η φίλη μου, η κυρία Βρεζιά, μίλησε για ένα θέμα που δεν ήθελα να φυγεί σήμερα. Δυστυχώς, η Τινησία έχει τρία, ένα τριπρό πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα στα νότια οι γειτονικέ μα χώρε, το είπατε, μιλήσατε και για τη Λιβύη μαζί με την Τινησία, αλλά από τι αρχέ του Δεκέμβρη υπάρχει ένα αρνητική ερνητικός κατάλογος ε, για... έχει καταχωριστεί στον κατάλογο των φορολογικών παραδείσων η... την Ισία. Είναι παράδεισος αλλά όχι φορολογικός πάντως. Ε, και σε κάθε περίπτωση λίγες μέρες μετά από την απόφαση αυτή ε, βγήκαμε και σε άλλο κατάλογο για λεύκανση παρανόμων προσόδων για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στην Τινησία από το 2011 Δυστυχώ, αντιμετωπίζουμε αυτό το νέο για μα φαινόμενο, την τρομοκρατία, τότε που δεν γνωρίζαμε καν τα όπλα, τα ναρκωτικά, την, ε, ε, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, τη διακίνηση ανθρώπων, η κατάσταση έχει εξελιχθεί αρνητικά. Και έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτά τα προβλήματα. Το να περιλαμβάνεται την Ισία σε αυτόν τον κατάλογο, τον αρνητικό, εμάς μας σώκαρε ήταν κόλαφος. Και θα θέλαμε να δοθεί χρόνο στην Τινησία για να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι και στο σωστό δρόμο είμαστε και ότι έχουμε προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Ξέρετε, οι βουλευτές στην Τινησία δεν έχουν γραφεία και ε, βοηθούς και έχουν και μια στίβα από φακέλους και δοσιά που πρέπει να εξετάσουν για να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να τους δώσετε και λίγο χρόνο για να μπορέσουν να εξηγήσουν, να επιχειρηματολογήσουν, να παρουσιάσουν ολοκληρωμένη την προσέγγισή μας. Για τον κατάλογο τώρα αυτό, τον μαύρο ή αρνητικό κατάλογο, ελπίζουμε, διότι η επιστολή των πολιτικών έφτασε κάπως καθυστερημένα, δεν προλάβαμε, αλλά το να περιληφθούμε σε αρνητικό κατάλογο κάπως μας ξαφνιάζει. Δεν μπορούμε παρά να είμαστε σοκαρισμένοι. Υπάρχουν χώρε που έχουν αναγνωριστεί από το Ευρωκοινοβούλιο ω φορολογική παράδειση και δεν έχουν περιληφθεί από τον κατάλογο. Ενώ η Τινησία, που από το 1962 έχει νομοθεσία για να ενθαρρύνει τι ξένε επενδύσει στη χώρα. Τι εργαλείο χρησιμοποιεί βάσει τη νομοθεσία τη. Έναν εικονικό φόρο για τι εταιρείε που θέλουν να επενδύσουν στην Τινησία. Είναι ο μόνο τρόπο που εντοπίσαμε από το 1972 για να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Και ξέρετε ότι τις χρειαζόμαστε ε, απελπισμένα, διότι έχουμε μία ενδημούσα ανεργία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί, 15% του πληθυσμού των νέων ιδιαιτέρως και μάλιστα των πτυχιούχων ε, της ανώτατης εκπαίδευσης. 650.000 ε, νέους άνεργους έχουμε και οι περισσότεροι είναι πτυχιούχοι. Έχω μια εικόνα που με... Ακόμα με προκαλεί δυσαρέστα συναισθήματα. Ένα άνθρωπο από την Υπεθρό που ε, κραδένει τα πτυχία των τέσσερων, των τεσσάρων παιδιών του, οι οποίοι όλοι πήγαν ε, πανεπιστήμιο και είναι όλοι άνεργοι. Ε, το οι προσπάθειές μας λοιπόν να ενισχύσουμε το κοινωνικό μας σύστημα έχουν καταλήξει στο να έχουμε βλάβη αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό έλεγα ότι έχουμε το πρόβλημα στην αρχή. Τις γειτονικέ χώρες το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο και τη χρηματοδότηση τη δημοκρατία που τώρα μα φορτώνεται, ε, Ποιο μπορεί να λέει ότι την Ισία χρηματοδοτεί την τρομοκρατία. Εμεί είμαστε σε διαρκή πόλεμο. Την προσπάθεια καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Και τώρα μα βάζετε σε ένα κατάλογο ξεπλήματο βρώμικου χρήματο και χρηματοδότηση και φορολογικών παραδείσων. Κάτι που πραγματικά ξαφνιάζει. Και ακούμε τόσα λόγια ενθάρρυνση από την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικώ και ο ιδιαίτερως από την πλευρά των Ευρωβουλευτών και ταυτόχρονα πέφτει ο Πέλεκης. Έπεσε πολύ η βαθμολογία της Τινησίας τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον κατάλογο θα ε, ασκηθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση στην ε, την ε, οικονομία και θα πληγεί και η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, η απασχόληση, η παραγωγή πλούτου. Ευχαριστώ και αν επιτρέπετε να δώσω και το λόγο στους υπουργού. Ευχαριστώ. Α, μια στιγμή, μια στιγμή λέει ο Πρόεδρος. Δεν είχαμε προγραμματίσει εκτενή συζήτηση για το θέμα αυτό. Και δεν έχουμε χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, μόνο χάρη να βρώτε, θα σας δώσω ένα λεπτό το λόγο. Αν και ξέρω τι θα πείτε. Θα είναι θετική απάντηση. Ένα λεπτό μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήρθα απλώ για να σα απευθύνω χαιρετισμό στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, γιατί είχα το προνόμιο και τη τιμή να σας υποδεχτώ εγώ στην Τινησία και διαπιστώνω με χαρά ότι ε, εκτιμήσετε ιδιαίτερο στην πρόσβαση που σας δώσαμε και την ευκαιρία να θέσετε τις ερωτήσεις σας και να λάβετε από πρώτο χέρι τις πληροφορίες που χρειαζόσασταν. Και μια και είμαι εδώ στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, θα ήθελα να σας πω ότι η Τινησία που ε, συγκροτείται μέρα με τη μέρα σε μια δημοκρατική διαδικασία, θα ήθελα ακριβώ ε, να ε, συνδεθεί με το ευρωπαϊκό μοντέλο και να αγκιστρωθεί εκεί, γιατί για, για μας είστε ένα μοντέλο και ένας χώρος ελευθερίας, παράδειγμα προς και πολύ σημαντικός. Και θέλουμε φυσικά προνομιακές σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς και το γεγονός ότι έχουμε έρθει ολόκληρη αντιπροσωπεία και με τον Υφυπουργό Εξωτερικού Εμπορίου που είναι ο ε, επικεφαλής της διαπραγμάτευσης για την ΑΛΕΚΑ. Ε, φυσικά θα συνεχίσουμε να συζητούμε και να απαντάμε σε ερωτήσεις στα πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων για αυτή τη συμφωνία. Και θέλω να δώσετε χρόνο στην Τινησία για να δημιουργήσει, να οικοδομήσει, να συγκροτήσει τη δημοκρατία της και να μην κολλήσει αυτή τη διαδικασία σε κάποια τεχνικά ή διαδικαστικά ζητήματα και να πληγεί από μια τέτοια με τέτοιο γραφειοκρατικό ή διαδικαστικό πρόσκομα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο και σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Κύριε Πρέσβη, η κυρία Βερζιά... Έφερε ακριβώ αυτό το θέμα της πέμπτης οδηγίας ε, περί ξεπλήματος χρήματος και δικαίω το έθεσε γιατί κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών ήρθαμε σε επαφή με την πρεσβεία γιατί προφανώς η Τινησία ήταν στον κατάλογο και αντιλαμβανόμαστε το παράδοξο, την ανησυχία που δημιουργείται. Και νομίζω το εξέφρασε πολύ σωστά η κυρία Βερζιά. Να εξηγήσω στους συναδέλφους το τι κάναμε εμείς, ότι απλώς η εν λόγω οδηγία δεν αφορά μόνο την Επιτροπή μας, αφορά και την Επιτροπή Οικονομικών. Πρόκειται περί κοινής αρμοδιότητας και, και οι δύο πρόεδροι των Επιτροπών επέκτηναν την προθεσμία για τις συζητήσεις για το θέμα της ε, Τινησίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές που κινήθηκαν τόσο γρήγορα. Ε, πρόκειται για ένα πρακτικό ζήτημα εμείς δηλαδή επισκεφθήκαμε την, την Ισία, αντιλαφθήκαμε την μεταναστευτική πίεση που αντιμετωπίζει η χώρα από πολλές πλευρές και βέβαια πρέπει να μιλήσουμε για μια πραγματική εταιρική σχέση και το γνωρίζουμε. Οπότε δράσαμε ταχύτατα και εκτιμούμε ιδιαιτέρως την συνεργασία. Τώρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο βήμα. Να χρησιμοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε δηλαδή για να αναπτύξουμε τα επιχειρηματά μας και θα είμαστε νομίζω σε στενή συνεργασία για να δούμε αν μπορεί να επιτευχθεί κάποια πρόοδος. Κάτι το οποίο οπωσδήποτε ενίσχυσε η σημερινή σας παρέμβαση. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Τώρα θα... Ε, ναι, το εξηγήσω στους συναδέλφους που δεν είχαν παρακολουθήσει το θέμα αυτό για τα ζητήματα ξεπλήματος χρήματος. Σας ευχαριστώ λοιπόν κύριε Πρέσβη. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι, περνάμε τώρα. Α, με συγχωρείτε. Ε, θα ήθελα να πω κάτι μεταξύ των δύο θεμάτων επί της διαδικασίας πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα αν μου επιτρέπετε επί της διαδικασίας συνειδητοποιώ πως για ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι και ο λόγος είναι ότι πολλοί πάμε και στην Επιτροπή Τρομοκρατίας που συνεδριάζει αυτή τη στιγμή και θα ήθελα να το επισημάνω στην γραμματεία της Επιτροπής, της δικής μας και της άλλης Επιτροπής, να διασφαλίσει ότι ειδικά Δευτέρα απόγευμα, όταν είναι ούτως ή άλλως τόσοι λίγοι συνάδελφοι παρόντες, να μην έχουμε δύο ταυτόχρονες συνεδριάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μετσόλα. Προσπαθούμε, προσπαθούν οι δύο γραμματείες να το συντονίσουν. Ε, δυστυχώς ένα από τα προβλήματα το να έχουμε μια ειδική επιτροπή όπου έχει παρόμοια στελέχωση αρκετοί βουλευτές είναι μέλη και στις δύο επιτροπές σημαίνει ότι θα υπάρξουν και κάποιες συνεδριάσεις που συμπίπτουν. Και εγώ είμαι μέλος στην ε, Επιτροπή για την Τρομοκρατία και η γραμματεία θα έχει φτάσει στα όρια της. Δυστυχώς έχουμε πολλά προβλήματα. Προσπαθούμε να τα συμβιβάσουμε, αλλά δεν θέλω να σας δώσω φρούδες ελπίδες ότι θα γίνει κάτι σύντομα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, εν πάση για να μην συμπίπτουν οι συνεδριάσεις. Και δεν είναι αυτός ο, ο μόνος λόγος για την χαμηλή προσέλευση των συναδέλφων, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Περνάμε τώρα στο σημείο 5. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5. Μια σημαντική ανταλλαγή απόψεων που είχαμε ζητήσει εμείς για την συνεισφορά της ε, Κομισιόν για την θεματική συζήτηση σχετικά με μια μελλοντική πορεία όσον αφορά την εξωτερική και εσωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής. Τον Δεκέμβριο δημοσιεύθηκε αυτή η ανακοίνωση, η οποία περιλαμβάνει διάφορα παραρτήματα σε ζητήματα τα οποία συζητούμε στην Επιτροπή μας για την επανεγκατάσταση και την δήλωση με την Τουρκία. Καλύπτει λοιπόν και την τρέχουσα κατάσταση στην εφαρμογή του νομοθετικού πακέτου για τη μεταρρύθμιση του Κοινοευρωπαϊκού συστήματο Ασύλου. Χαιρετίζουμε λοιπόν την δυνατότητα να δούμε τα ζητήματα αυτά υπό ένα ευρύτερο πρίσμα όπως είχαμε ήδη προτείνει στην έκθεσή μας για την κατάσταση στη Μεσόγειο και μια ολιστική αντιμετώπιση της ε, μετανάστευσης, της εκθέσεις ε, Μετσόλα και Κιέγγε. Οπότε τώρα θα θέλουμε να ακούσουμε πώς ε, πηγαίνουν τα πράγματα από τον Σάιμον Μόρντιο, ο οποίος προσφέρθηκε να μας ενημερώσει και είναι αναπληρωτής ε, γενικός ε, διευθυντής ε, της σχετικής διεύθυνσης αυτής και θα ακούσουμε μετά και έναν εκπρόσωπο της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Αγαπητέ Σάιμον, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. καλή χρονιά σε όλους, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε με την ανακοίνωση αυτή της 7ης Δεκεμβρίου είναι να καθορίσουμε έναν ξεκάθαρο οδικό χάρτη με κάποιες δράσεις κλειδιά που θα μας βοηθήσουν να πετύχουμε μια γενικότερη, ένα γενικότερο συμβιβασμό που θα περιλαμβάνει, ελπίζουμε, και απτή προόδο στο σύστημα ασύλου. Πριν περάσουμε στην ουσία, Να σας δώσω κάποια νούμερα. Βλέπουμε από τους αριθμούς ότι υπάρχει κάποια πρόοδος στις αρχές του 2018, τους τελευταίους 12 μήνες. Παραδείγματος βλέπουμε ότι ο αριθμός των ανθρώπων που χάνονται στην Μεσόγειο έχει μειωθεί από γύρω στα 4.000 άτομα το 2016 σε 2.832 το 2017. Βεβαίως εξακολουθούν να είναι 2.800 άτομα παραπάνω από όσο θα έπρεπε, αλλά ο αριθμός μειώνεται. και βεβαίως ε, έχουμε τις αφήξεις που έπεσαν στην Ελλάδα το 2017 στις 35.000 από 177.000 ε, το 2016. Επίσης είχαμε μια δύσκολη αρχή του 2017 και μια σημαντική μείωση των αφήξεων στην Ιταλία από 180.000 το 2016 σε 119.000 το 2017 μία μείωση κατά 30% για την πλευρά της προστασίας νομίζω ότι είδαμε δύο επιτυχή προγράμματα επαναγκατάστασης ε, πάνω από 25.000 ευπαθή άτομα πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν δείτε τα συνολικά νούμερα Μιλάμε για 80.000 άτομα παγκοσμίω, ε, μιλάμε για μεγάλη αλλαγή πλέον και περνάμε σε μια φάση ε, μετεγκατάστασης και είχαμε γύρω στα 33.000 άτομα ε, που έχουν υποβάλει αίτηση μετεγκατάστασης από την Ελλάδα. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα γιατί βεβαίως απασχολεί πολύ τον τύπο το ζήτημα. Αυτό το οποίο προσπαθούμε εμείς να περάσουμε ως βασικό μήνυμα στην ανακοίνωση είναι ότι υπάρχει πρόοδος, αλλά χρειάζεται ακόμα ε, δουλειά σε όλα αυτά τα μέτωπα, σε όλες αυτές τις δράσεις και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικέ προκλήσεις και να μην έχουμε μόνο λύσεις ad hoc που είχαν βεβαίως αποτελέσματα ε, και γνωρίζω πως είναι κάτι το οποίο ζητάει και το Κοινοβούλιο. Το έχουμε συζητήσει ε, πολλές φορές και θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με έναν τρόπο συνολικό στην εσωτερική και την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής αλλιώς δεν θα έχουμε ένα συνολικό σύστημα το οποίο θα επιτέχει μια ισορροπία μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποιο μαγικό μέτρο το οποίο θα μας δώσει μια απάντηση από μόνο του. Γιατί υπάρχει μια πολύπλευρη ε, κατάσταση και νομίζω ότι θα επιτύχουμε φέτος και μακροπρόθεσμα εάν ε, σημειωθεί πρόοδο σε όλα τα μέτωπα. Να πω τώρα λίγα λόγια για τα βασικά μηνύματα της άνωσης για τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου. Έχουμε υποβάλει τις σχετικές προτάσεις το 2016 και νομίζω πως έχει φτάσει η στιγμή να επιτύχουμε μια συμφωνία. Έχουμε έναν οδικό χάρτη που έχουμε υποβάλει που θα μας επιτρέψει μέχρι τα μέσα του 2018 να έχουμε απτή πρόοδο. Ελπίζουμε να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια αίσθηση του κατεπήγοντος τουλάχιστον στο Συμβούλιο Πρέπει λοιπόν να μην λειτουργούμε μόνο υπό καθεστώς ε, και πίεση κρίσεως ε, και βεβαίως αυτό δεν θα γινόταν αν υπήρχε ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Θα πρέπει λοιπόν ε, οι συνομοθέτες να φροντίσουν ο βασικός στόχος να είναι η μεγαλύτερη σύγκληση και να καταπολεμήσουμε τα κίνητρα για δευτερογενείς μετακινήσεις. Θα πρέπει να προσφέρουμε καλύτερη και γρηγορότερη προστασία σε αυτούς οι οποίοι την χρειάζονται, αλλά ταυτόχρονα να μην επιτρέψουμε την κατάχρηση του συστήματος και να επιστρέφονται τα άτομα τα οποία δεν δικαιούνται προστασία. Πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε κάποιες κοινέ ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ε, κάτι το οποίο προσπαθούμε και από ό,τι φαίνεται συχνά δεν γίνεται αντιληπτή η κοινή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα σχετικά θέματα. Υπάρχει και ο Πίτερ Νίντερμαϊρ εδώ. Έχουμε συνεργαστεί και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου. Έχουμε επιτύχει μια συνολική συμφωνία. Βλέπουμε σταθερή πρόοδο στο σύστημα δακτυλικών αποτυπωμάτων, το Eurodac, αλλά συνεχίζεται η πρόοδος ε, στον ε, κανονισμό περί προϋποθέσεων, ε, στις συνθήκες υποδοχής, ε, στον κανονισμό διαδικασιών ασύλου. Ε, χρειάζεται ακόμα δουλειά και από την πλευρά του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνομοθετών να ξεκινήσουν, ελπίζουμε τον Μάιο. Τώρα, τέλος, να στραφώ στο θέμα του Δουβλίνου. Δεν νομίζω ότι καμία μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου μπορεί να επιτύχει χωρίς ε, ε, μια μεταρρύθμιση του συστήματος για να μοιραστούμε την ευθύνη και την αλληλεγγύη. Γνωρίζουμε πως εδώ πέρα κλειδί είναι η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου και η μόνη ε, σωστή λύση για το μέλλον. Εσείς ως κοινοβούλιο έχετε ήδη εγκρίνει την θέση σας, είναι σαφής και έχει φτάσει η στιγμή νομίζω να καταλήξουν σε μια κοινή θέση και τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι η Βουλγαρική Προεδρία έχει εμπλακεί, έχουμε μια νέα όρμη στις διαπραγματεύσεις, έχει ήδη συνεδριάσει η ομάδα εργασίας, θα συνεδριάσει με συγχωρείτε αυτή την εβδομάδα. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία επίσης να επαναλάβω κάποια μηνύματα που ανέφερε εντόνως ο επίτροπος στο Κοινοβούλιο. Δεν θεωρώ πως η μεταρρύθμιση του Δουβλίνου χωρίς ένα στοιχείο μετεγκατάστασης, ειδικά για καταστάσεις κρίσης, ε, θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε σε μελλοντικές κρίσεις. Και θα είμαι σαφής. Κάποιοι προσπάθησαν να πούν ότι ε, απέτυχε η μετεγκατάσταση. Ε, δεν συμφωνώ. Αν το δούμε ουδέτερα και αντικειμενικά, θα δούμε ότι είναι ένα επιτυχές μέσο στήριξης της Ελλάδας και της Ιταλίας και βοηθάει τον κόσμο να έχει πρόσβαση στα δικαιώματά του και νομίζω ότι αν δει κανεί τα στατιστικά στοιχεία είχαμε γύρω στα 35.235 άτομα τα οποία ήταν επιλέξιμα για μετεγκατάσταση και 33.000 ε, σχεδόν ε, μετεγκαταστάθηκαν. Τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για ένα ποσοστό εφαρμογής 93%. Ναι, είμαι σαφής. Ε, δεν έχει σταματήσει η ανάγκη μεταγκατάστασης και νομίζω πως θα πρέπει όσο περιμένουμε να εφαρμοστεί το Δουβλίνο κάτι το οποίο είναι επίγον θα πρέπει τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη και εμείς θα φροντίσουμε να υπάρξει οικονομική στήριξη. Αλλά παράλληλα με αυτό να τονίσω ότι θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε όλους τους άλλους πυλώνες ε, μια συνολικότερης προσέγγισης ε, της μετανάστευσης και να αναφέρω κάποια από αυτά τα βήματα. Πρώτα απ' όλα να προστατευτούν τα εξωτερικά μας σύνορα. Έχει περάσει 1,5 έτος από την ε, εντολή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Συνοριοφυλακής και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε πλήρως. Η υπηρεσία προχωρά. Βλέπουμε ότι έχει αναπτύξει 1.700 σύνοριοφύλακες, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα και νομίζω ότι μέχρι τον Μάρτιο πρέπει η συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή να έχει το υλικό και το προσωπικό που απαιτείται ξεκολουθούμε να υστερούμε. Γύρω στα 200 άτομα λείπουν για την δύναμη ταχεία αντίδρασης. Ε, μόνο 14 ε, κράτη-μέλη έχουν συνεισφέρει στο υλικό. Δεν επαρκεί αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσετε κι εσείς την πίεση και σημαντικό είναι να υπάρξει μια αύξηση των επιστροφών και εγώ έχω δεσμευτεί ότι θα σας ενημερώνω για να γνωρίζετε. Ξέρω πως είναι επίμαχο ζήτημα, αλλά είμαστε υπέρ της πλήρους διαφάνειας και κάτι το οποίο πρέπει να γίνει εδώ πέρα είναι ένα τεράστιο άλμα αύξησης των επιστροφών που κάνουν και τα κρατημέλη και η σχετική η κοινοτική υπηρεσία και τον Δεκέμβριο είχαμε θέσει φιλόδοξους στόχους. Είπαμε ότι θα θέλαμε να επιτύχουμε μια αύξηση 30% μέχρι το Μάρτιο και 50% μέχρι τον Ιούνιο του 2018 επίσης. Θέλουμε να γίνουν πολύ περισσότερα για τις νόμιμες διόδους, να υπάρχουν επαρκείς νόμιμες δίωδοι. Θα θυμάστε ίσως πως ζητήσαμε τον Σεπτέμβριο από τα κράτη-μέλη να επαναγκαταστήσουν τουλάχιστον 50.000 άτομα μέχρι το τέλος του 2019. Τα καλά νέα είναι ότι ήδη έχουμε λάβει πολύ συγκεκριμένες ε, δεσμεύσεις, 40.000 ε, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον στόχο των 50.000 και πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα στην ε, νόμιμη οικονομική μετανάστευση για να δούμε κάποιες προκλήσεις που αφορούν και το εργατικό δυναμικό και συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για να δούμε τα πρώτα έργα για κάποιες συγκεκριμένες χώρες εταίρους για την νόμιμη οικονομική μετανάστευση και βεβαίως σημαντικό είναι ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, κατέληξαν σε συμφωνία για την μπλε κάρτα που θα μας επιτρέψει να προσελκύσουμε οι άτομα υψηλής εξειδίκευσης. Ε, και τέλος, ο κύριος Νικόλοφ εδώ πέρα, ο συνάδελφος από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, θα πει κάποια πράγματα. Και έχουμε βεβαίω και την δήλωση για την Τουρκία και θα δούμε τι θα γίνει με την κατάσταση στη Λιβύη. Σκοπεύω και εγώ να ταξιδέψω τις επόμενες ημέρες ε, στη Λιβύη με τους ε, συναδέλφους ε, για να δούμε το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί. Βλέπουμε μια σημαντική αύξηση στις εθελοντικές επιστροφές και ελπίζουμε μέχρι τον Φεβρουάριο να δούμε άλλες 50.000 εθελοντικές επιστροφές από την Λιβύη και βλέπουμε τις πρώτες εκενώσεις από την Λιβύη προς τον Νίγηρα και μετά κάποια μετεγκατάσταση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν να έχουμε κάποια μετεγκατάσταση μέχρι τον τέλος Φεβρουαρίου. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να τονίσω, που είναι σημαντικό, θέλουμε τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν στα ταμεία τα οποία προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις αιτίε μετανάστευσης, ειδικά στην Βόρεια Αφρική υπάρχει έλλειψη 340 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε θα ήθελα να επαναλάβω κάποια πράγματα. Ότι τώρα πρέπει να φύγουμε από την αντίδραση ad hoc σε μια δομημένη αντίδραση. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα ένα, ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και επιπλέον πρέπει να εργαστούμε και στα άλλα μέτωπα γιατί αυτή η διασύνδεση είναι το κλειδί για να μπορούμε να έχουμε ε, μια επιτυχή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου. Ευχαριστώ. Very much, Simon. Σε ευχαριστούμε, Σάιμον. Ο κύριο Νικόλοφ τώρα από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που αντικαθιστά την κυρία Λότε Κνούτσεν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να στήσω συγγνώμη εκ μέρους κυρία κυρίας Κνούτσεν που κολλείται σήμερα. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω δύο συγκεκριμένα θέματα σε ό,τι αφορά την πρόοδο που υλοποίησαμε στην συνεισφορά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις εξωτερικές πτυχές, στην εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Έχουμε σημειώσει κάποια πρόοδο στο διάδρομο της Κεντρικής Μεσογείου και το δεύτερο συναφές θέμα αφορά την κατάσταση της συζήτησης ε, ε, της παγκόσμιας συζήτηση για τη μετανάστευση. Εμείς τις τελευταίες δύο εβδομάδες επικεντρωθήκαμε ιδιαίτερα στο θέμα της, του διαδρόμου της Κεντρικής Μεσογείου και προσπαθήσαμε να θέσουμε σε εφαρμογή την τριμερή ε, ομάδα κρούσης που ξεκίνησε στις 13 Νοεμβρίου μετά την ε, Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική και προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των μεταναστών από τη Λιβύη και μάλιστα καταφέραμε οι εταίροι μας από την Αφρικανική Ένωση αλλά και οι εταίροι μας από τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και ο Οργανισμός για τους Πρόσφυγες ε, του ΟΗΕ να συνεργαστούμε. Είχαμε πολυάριθμες συναντήσεις και σε επιχειρησιακό επίπεδο στην Μπέμπα και σε πολιτικό επίπεδο εδώ στις Βρυξέλλες παρουσία της είπα της εκπροσώπου στις 14 Δεκεμβρίου και μία επίση συνάντηση που κάναμε στην Τινησία λίγο πριν τις διακοπές ε, στην Τίνιδα με τον πρέσβη μας και εκπροσώπους της Αφρικανικής Ένωσης ε, και παρουσία εκπροσώπων των δύο οργανισμών. Όπως είπε ο κύριος Σάιμον Μόρντιου, ε, προετοιμάζουμε και την ομάδα υψηλού επίπεδου για την επίσκεψη που θα πραγματοποιήσει στα τέλη του μήνα στην Τρίπολη. Ένα σημαντικό ζήτημα που θα ήθελα να τονίσω είναι ο συνεχής και δέλτος συντονισμός που έχουμε με τις λιβικές αρχές. Κρατούμε αδιάλειπτες αυτές τις επαφές και το συντονισμό, ώστε η συνεργασία και σε πολιτικό και σε επιχειρησιακό επίπεδο να είναι εξασφαλισμένη και αυτός είναι και ο σκοπός της επερχόμενης ε, επίσκεψης υψηλού επίπεδου. Σε ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, ένα από αυτά είναι το θέμα της πρόσβασης στα κέντρα υποδοχής ε, της ε, Λιβύης. Αυτό μέχρι στιγμής ήταν το πιο προβληματικό ζήτημα. Πάντως, κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε συνεργασία με τις Λιβύικες Αρχές και με τους οργανισμούς ε, του, ε, των Ηνωμένων Εθνών, να εξασφαλίσουμε παρουσία της Παγκόσμιας Οργάνωσης για τη Μετανάστευση και της για τους πρόσφυγες ε, στα κέντρα κράτησης και να εξασφαλιστεί η προστασία των μεταναστών με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Το δεύτερο ζήτημα που επίσης μας απασχολεί είναι η πρόβλεψη της προξενικής βοήθειας ώστε να, να μπορέσουμε να επαναπατρίσουμε ε, χωρίς προβλήματα τους μετανάστες και σε αυτό υπολογίζουμε και στη συνεργασία με τους εταίρους μας από την Αφρικανική Ένωση που μας βοηθούν για να εξασφαλίσουμε τέτοια προξενική ε, υποστήριξη στις χώρες της Αφρικανικής Ένωσης κυρίως και ιδίως εκεί που δεν έχουμε μόνιμα προξενία όπως στη Λιβύη ή ε, μάλλον σε χώρες που δεν έχουν μόνιμα προξενία στη Λιβύη. Επίσης, ε, σημειώνουμε πρόοδο στα προγράμματα επανένταξης στις χώρες προέλευσης μετά την ε, επιστροφή των μεταναστών στις πατρίδες τους. Και μέχρι τα τέλη του έτους, με βάση τις πληροφορίες που μας δίνει η Διεθνής Οργάνωση για τη Μετανάστευση, είχαμε περίπου 20.000 ε, οικειοθελείς επιστροφές ε, για όλο το χρόνο στη Λιβύη με παροχή βοήθειας, τεράστια αύξηση δηλαδή σε σχέση με τις χίλιες περίπου οικειοθελείς επιστροφές με υποστήριξη που είχαμε πέρυσι. Φέτος 20 ε, ο αριθμός. Και σε συνεργασία που είχαμε όχι μόνο με το, τους οργανισμούς τους φορείς των Ηνωμένων αλλά και με την Αφρικανική Ένωση ε, καταφέραμε να εντοπίσουμε την ανάγκη να αντιμετωπίσουμε πιο σφαιρικά τις ε, μεταναστευτικές προκλήσεις και αντιληφθήκαμε ότι χρειάζεται μια πιο ε, δραστήρια συμπεριφορά και από τους εταίρους μας Αφρικής για την υλοποίηση αυτού του στόχου. Έτσι ενισχύσαμε και διαβρύαμε τις συζητήσεις ε, που έχουμε εμείς με τους Αφρικανούς εταίρους και σε παγκόσμιο επίπεδο για να δοκιμάσουμε και εμπράκτος ε, την διυπηρωτική συνεργασία. Κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι απαραίτητο και σημαντικό για τις τρέχουσες συζητήσεις για τα δύο παγκόσμια σύμφωνα για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες ε, που βρίσκονται εν εξέλιξη. Και επίσης ε, ετοιμάζουμε τις επίσημες διαπραγματεύσεις για το Παγκόσμιο, για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση που θα ξεκινήσουν ε, τις, τον επόμενο μήνα με βάση το σχέδιο που περιμένουμε για τα τέλη του μήνα. Και προετοιμάζουμε τη δική μας στάση ε, και θέση για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Αυτό που ήθελα να τονίσω είναι η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, καθ' όλη τη διάρκεια του 2017 να αποφαίνεται με ενιαία φωνή. Αυτή η ομοφωνία και η ομόνοια ήταν πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα όλες οι χώρες ομόφωνα συμφώνησαν για την συμμετοχή μας στην παγκόσμια αυτή συζήτηση και στις θέσεις που θα προβάλλουμε και θα υποστηρίξουμε στις ε, παγκόσμιες διαπραγματεύσεις για το σύμφωνο αυτό για τη μετανάστευση. Μέχρι στιγμής πάντως αυτή η σύμπνοια ήταν ευπρόσδεκτη και τα αποτελέσματα έδωσαν μια ομόφωνη θέση όλων των κρατών μελών στην προπαρασκευαστική φάση των διαπραγματεύσεων. Κάτι που προϊονίζεται καλή προετοιμασία και για το αποφασιστικό τμήμα των διαπραγματεύσεων που θα λάβει χώρα στη διάρκεια του 2018. Ελπίζω να συνεχιστούν οι συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και στη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας και να συνεχιστεί η αγαστή συνεργασία μας ώστε να συνεχιστεί αυτή η ομόφωνη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ερχόμενες φάσεις των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Απευθείας πάμε στους βουλευτές και στη σειρά με την οποία ζήτησαν το λόγο, κυρία Κιέγγε. Δύο λεπτά αν μπορείτε όλοι. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Κλοντ. Μερικές παρατηρήσεις θέλω να κάνω, διότι η σημερινή συζήτηση έχει ως αφετηρία και την παρακολούθηση, την αξιολόγηση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της κυρίας Μετσόλα και το δικό μου. Εκεί θέλαμε μια ολιστική προσέγγιση για να σταματήσουμε να έχουμε την ε, συγκυριακή προσέγγιση που επί χρόνια επικρατούσε. Χρειάζονται νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, διότι αν θέλουμε να ξεφύγουμε από την αντιμετώπιση απλώς επιβουσών καταστάσεων και να έχουμε μια προσέγγιση μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, πρέπει πάνω απ' όλα να επενδύσουμε σε νομοθετικά εργαλεία. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημείο αφετηρίας. Και ένα από τα βασικά σημεία του εγγράφου μας αφορούσε την αλληλεγγύη. Ξεκινώντας από το γεγονός ότι βεβαίως χρειάζεται και διάσωση, η διάσωση ανθρώπινων ζώων. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό για μας και να μην ξεχνάμε ότι και η 6η Ιανουαρίου φέτος είναι μια ημερομηνία που επιτρέπει σε εμά, στι περισσότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να γιορτάζουμε λιγότερες ε, απώλειες ανθρώπινων ζώων στη θάλασσα. Όμως αυτό δεν έχει πάυσει. Ήδη ε, στις 6 Ιανουαρίου 64 ανθρώπινες ζωές χάθηκαν, άρα η διάσωση συνεχίζει να είναι απαραίτητη. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τα νομοθετικά μας εργαλεία και να προχωρήσουμε στην μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Εύχομαι το Συμβούλιο και με τη νέα Βουλγαρική Προεδρία που τώρα ξεκινά να δείξουμε το απαραίτητο θάρρος, την τόλμη που έδειξε και το Κοινοβούλιο και να προχωρήσουν στην ε, μεταρρύθμιση του Δουβλίνου, ώστε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες που τον αλογούν. Ολοκληρώνοντας, να πω ένα σημείο, να αναφέρω ένα σημείο που δεν μου είναι πολύ σαφές, διαβάζοντας ε, το έγγραφο που και εσείς μας παρουσιάσατε. Ένα σημείο που μιλά για ε, επαρκή ένδικα μέσα λέγοντας ότι μέχρι τώρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε, έχουμε χρησιμοποιήσει τη γαλάζια κάρτα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να δώσουμε δυνατότητες νομίμης μετανάστευσης μέχρι το Μάρτιο του 2018 στις χώρες εταίρους μας. Γιατί ακριβώς μιλάτε και μπορείτε να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιο θα είναι αυτός ο δικός χάρτης και για το, όσα προέκυψαν από τη Σύνοδο του Αμπιτζάν για την διαχείριση των σχέσεων μας με τη Λιβύη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ με Σεσίλ, ο κύριος Νίντερμιλερ. Ευχαριστώ. Καταρχάς σας ευχαριστώ και τους δυο για τις παρουσιάσεις σας. Μιλήσατε πολύ για σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Καλό είναι να τη βλέπουμε για αυτή την πρόοδο, αλλά επιτρέψτε μου να μιλήσω περισσότερο για τα προβλήματα που έχουμε ακόμη. Πρώτα απ' όλα είμαι απολύτως βέβαιος ότι το θέμα της μετανάστευση, το θέμα των προσφύγων, είναι μείζονο σημασία, ε, θα είναι μείζονο σημασία και το 2018 όπως και τις προηγούμενες χρονίε. Σημαντικό λοιπόν είναι αυτό που αναφέρατε, ότι είναι η τέλεια συγκυρία για να κάνουμε κάτι περισσότερο. Και να δημιουργήσουμε ένα κοινό, ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Ταυτόχρονα όμω οφείλω να πω ότι είναι ξεκάθαρο πώς το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή, αλλά κυρίως το Συμβούλιο, χρησιμοποιούν διαφορετικούς ε, τρόπους να εκφραστούν για το θέμα και διαφορετικές μεθόδους. Δεν γίνεται ε, μία κάθε Προεδρία μάλλον βάλει την λήψη απόφαση στην επόμενη. Καμία Προεδρία και το Συμβούλιο το ίδιο δεν είχε την πολιτική τόλμη να λάβει μια πραγματική απόφαση. Και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο Ολοκληρώσαμε την εξέταση των δοσιέ που είχαμε στα χέρια μας τα τελευταία χρόνια και δεν είχε γίνει τίποτα στην πράξη. Δηλαδή και η Βουλγαρική Προεδρία θα πρέπει να δείξει το απαραίτητο ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Δεν ε, είναι κάτι που μπορούμε να το ανεχτούμε αυτό από το Ευρωκοινοβούλιο, αυτήν την αδράνεια. Κάτι άλλο τώρα. Αναφέρατε τον Οργανισμό για το Άσυλο. Φτάσαμε σε πολιτική συμφωνία το περασμένο καλοκαίρι. Για τους προηγούμενους έξι μήνες δεν έγινε τίποτα επί του θέματος. Το Συμβούλιο λέει ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Μα νομίζω είναι καθήκον του Συμβουλίου να δημιουργήσει τις συνθήκες για να υπάρξει συμφωνία. Ή, ε, λέει το Συμβούλιο χρειαζόμαστε μια συμβαστική λύση και να συμφωνήσουν και οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών. Και τι έχει γίνει, δεν υπάρχει καμία διάθεση για εξέβρεση συμβιβασμού από καμία πλευρά. Εάν συνεχίσουμε λοιπόν έτσι, θα έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα το 2018 από ό,τι το 2017. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να πω ότι βεβαίως εδώ έχουμε και έναν ελέφαντα στην αίθουσα, ο οποίος είναι η απουσία του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο δυστυχώς έχει πολύ κακή, ε, κακό ιστορικό στο θέμα αυτό, να το πω ε, προς όλους και το ίδιο έγινε και κατά τη διάρκεια του Χριστουγεννιάτικης Διακοπής βεβαίως. Η κυρία Σπινέλη, ευχαριστώ Πρόεδρε και καλή χρονιά. Πρέπει να πω ότι υπάρχει κάτι εδώ που δεν με πείθει τις εκφράσεις που χρησιμοποίησαν οι εκπρόσωποι της Επιτροπής είναι η τάση να παρουσιάζονται πολιτικές επαναπατρισμού και μείωση των αφήξεων στην Ευρώπη ως ε, δείγμα ανθρωπιστικής προόδου. Να εξηγήσω τι εννοώ. Εάν στην Ευρώπη φτάνουν λιγότεροι μετανάστες ή τέλος πάντων πρόκειται να ε, σταλούν πίσω στις χώρες τους, θα υπάρχουν λιγότεροι νεκροί. Αυτό δεν μου φαίνεται ολιστική προσέγγιση, μου φαίνεται σοφιστία. Ε, η δεύτερη ερώτησή μου αφορά τον επαναπατρισμό και τις ε, μετεγκαταστάσεις στην Λιβύη. Θέλουμε να εκενωθούν τα κέντρα κράτησης. Πολύ δύσκολο να γίνει πράξη αυτό. Πριν από τα Χριστούγεννα, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Κόστελ εξήγησε ότι είναι σχεδόν αδύνατο να έχει κανείς πρόσβαση σε μια σειρά από κέντρα κράτησης, ακριβώς γιατί δεν ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται. Και ότι έτσι κι αλλιώς, εφόσον εκενωθούν, την ίδια στιγμή ξαναγεμίζουν. Σε ό,τι αφορά ε, την μετανάστευση και τη γαλάζια κάρτα, και εδώ η δική μου η άποψη είναι λιγότερο αισιόδοξη από τους εκπροσώπους της Επιτροπής για την επανεγκατάσταση, την με την κατάσταση Το να το παρουσιάζουμε αυτό ως ε, αποτελεσματικό εργαλείο και να μιλάμε για φιλόδοξη γαλάζια καρτά νομίζω ότι είναι μια οφθαλμαπάτη και μια ψευδέστηση δεδομένη τη συμπεριφορά του Συμβουλίου. Και μετά σε ό,τι αφορά τι θεωρητικέ δεσμεύσει μα στο Νίγηρα. Ε, τι ακριβώ θεωρητική δέσμευση έχουμε αναλάβει. Διότι στην Ιταλία γίνεται πολλή κουβέντα για την αποστολή στρατιωτών από το Ιράκ στον Ιγυρά. Μπορείτε να μας πείτε τίποτα περισσότερο επί του θέματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μπάρμπαρα. Ρομπέρτα. Ευχαριστώ που ήρθατε και αφιερώνουμε χρόνο σε αυτό το σημαντικό θέμα. Μακάρι ήταν παρόν και το Συμβούλιο βέβαια για να απαντήσει τις απορίες του κυρίου Νίτερ Μίλλερ. Πάντως το Έλκιν είναι υπέρ ε, της ε, πρότασης ε, για τη μετανάστευση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι και λογική και διορατική, λαμβάνοντας υπόψη το πολύπτυχο χαρακτήρα του φαινομένου της μετανάστευσης. Έχουμε το πλαίσιο για τη μόνιμη επανεγκατάσταση που ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να βοηθήσουμε τους χρήζοντες βοήθεια ενώ εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες για να αποτρέψουμε την κατάχρηση του συστήματος. Χρειαζόμαστε νόμιμες, ε, νόμιμες μεθόδους ε, για να ε, αντιπαραδεχθούμε στα παράνομα κυκλώματα και συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης. Και ταυτόχρονα θέλουμε αυστηρές αλλά ανθρωπιστικές πρακτικές επιστροφών, ώστε να έχουμε πραγματικά διαδικασίες που θα καταλήγουν είτε σε ουσιαστική ενσωμάτωση είτε σε επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ένα μικρό ποσοστό έχει επαναπατριστεί και έχουμε περιλάβει και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και για το Μάλι, για παράδειγμα, το ποσοστό επιστροφών είναι 4,5%. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά επιστροφών. Θα πρέπει λοιπόν να αφιερώσουμε τους πόρους μας στους ε, πραγματικά αναξεπαθείς και χρήζοντες προστασίας. Επίσης, η πρόοδος μερικές φορές είναι εκνευριστικά αργή, αλλά κάποια πρόοδος υπάρχει, όπως με τη Γάμπια, το Μπαγκλαντές και το καθεξής. Και μάλιστα έχουμε ένα ε, γενναιόδωρο πακέτο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα χώρες προέλευσης και διέλευσης και βοηθήσαμε ε, στον αυληθούν ε, κάποιες από τις καταστροφικές ε, συνθήκες της Λιβύης. Αλλά για να είμαστε ειλικροί θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Επίσης, ε, το τρέχον πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο υποχρηματοδοτεί τα θέματα ασφάλεια και μετανάστευση. Θέλουμε ένα χρηματοδοτικό επίπεδο που θα ανταποκρίνεται στι πραγματικέ ανάγκε αυτών των τομέων και θα στηρίξουμε τι χώρε για να αντιμετωπίσουν τις ρίζες του φαινομένου της μετανάστευσης. Επίσης ε, θα πρέπει να έχουμε και χρηματοδότηση όχι μόνο των αναπτυξιακών ταμείων, αλλά να, να και τις ε, ευρωπαϊκές εταιρείες να αναπτύξουν σε αναπτυσσόμενες χώρες να επενδύσουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Και όταν έχουμε κάποιες εξαγγελίες να τις χρηματοδοτούμε και όλα. Κύριε Γκραπίνη, σας ευχαριστώ. Nu, Libe a pornit așa în forță cu o dezbatere extrem de interesantă. Η έναρξη τη κονιά με αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση είναι ένα πολύ καλό δείγμα. Ο κύριο Μορδιού έκανε μια πολύ αισιόδοξη παρουσίαση και πράγματι οι αριθμοί δείχνουν κάποιε ελαφρε βελτιώσει. Όμω στην ουσία του θέματο υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μα είναι σαφή. Κάποια από αυτά τα έθιξαν οι συνάδελφοι, εγώ ήθελα να προσθέσω κάποια ακόμη. Ε, για παράδειγμα, μπορείτε να μας πείτε αν όλα όσα υπόθηκαν για τη μεταρρύθμιση του συστήματος του ασύλου, τα νομοθετικά προβλήματα, μπορείτε να μας πείτε αν όλα εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο από τα κράτη-μέλη. Λέτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν με συγκεκριμένα κονδύλια. Εμείς έχουμε λάβει feedback και γνωρίζουμε ποια είναι η θέση των κατομελών στο Συμβούλιο, διότι εμείς στο Κοινοβούλιο λέμε αυτά που θέλουμε, το ίδιο και η Επιτροπή, αλλά το Συμβούλιο δεν κάνει τίποτα. Επίσης για, την, ε, ε για τις σχέσεις και τη συμφωνία με την Τουρκία. Ποια είναι η πρόπτικη της Επιτροπής για τις σχέσεις με την Τουρκία. Και τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με αυτό που είπε η προηγούμενη συνάδελφος, η κυρία Μετζόλα. Εφόσον γίνει αυτή η μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου, θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την προστασία, την ασφάλεια. Για την ώρα ε, έχουμε σαφείς διαδικασίες για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι οικονομικοί μετανάστες και ποιοι έρχονται από περιοχές με συγκρούσεις, ένοπλες συγκρούσεις. Ευχαριστούμε κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Μερικά από αυτά που ακούσαμε είναι ευπρόσδεκτα, αλλά καλύτερα τώρα να επικεντρωθούμε σε απορίες και ερωτήσεις. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σωστή η ισορροπία μεταξύ του προϋπολογισμού για το γραφείο για το άσυλο και των δυνάμεων κρούση, γιατί λέμε ότι το ΙΑΣΟ θα μετατραπεί σε ένα νέο οργανισμό. Οπότε η έμφαση που δίνεται στι επιστροφέ που δεν είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου, γιατί η, στο πακέτο αρχικά δεν περιλαμβανόταν και οι επιστροφέ. Τώρα παραδίνουμε ε, σημασία σε αυτό το θέμα. Υπάρχει όμω η επαρκή χρηματοδότηση ώστε το γραφείο αυτό να ανταπεξέλθει και στο ρόλο που έχει για το σύστημα ασύλου για να μην, για να μην ενισχύουμε την ευθύνη προς την Ελλάδα. Θα πρέπει λοιπόν να περικοδοτήσουμε και με τα το ΙΑΣΟ για να ανταπεξέλθει στο έργο του. Επίσης είπαμε ότι θα ε, αφήσουμε τις μεμονωμένες λύσεις και θα περάσουμε σε πιο συστημικές. Τι θα γίνει τότε με τη ρυθμίση με την Τουρκία θα έχουμε μια επισημοποίηση της ε, με συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συζήτηση ή θα συνεχίσουμε αυτές τις άτυπες ρυθμίσεις και διαθετήσεις αντί να τους δώσουμε ένα πιο καταστατικό και πιο συστημικό χαρακτήρα. Και όταν εννοώ καταστατικό ή κανονιστικό, εννοώ την πλήρη συμμετοχή και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, ε, αρχικά ακούσαμε κάποια σχόλια για τις μετακινήσεις ε, εκτός της Λιβύης. Καλό αυτό, αλλά με προβληματίζει αυτή η ρύθμιση με τη κυβέρνηση της Λιβύης, όποια και είναι αυτή. Επίσης, αυτές οι μετακινήσεις πώς θα ελεγχθούν, γιατί βλέπουμε στην Κάμπια τι γίνεται. Εκεί υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ αυτών που ακούν στη Λιβύη οι άνθρωποι αυτοί και το τι συναντούν όταν φτάνουν στην Κάμπια. Θα γίνει μια επαρκής παρακολούθηση αυτών των μετακινήσεων με ενημέρωση κατόπιν για τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ. Όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι ήδη, ε, δεν θα επανέλθω κι εγώ στην απουσία του Συμβουλίου, το είπαν οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό σε πολλές συζητήσεις πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς στο τι λέμε. Τα άτομα αυτά, τα οποία φεύγουν λόγω πολιτικών διώξεων, βασανιστήριων, πολέμου, έχουν δικαίωμα προστασίας κτλ. Αυτό είναι πέραν πάσης αμφισβήτησης, αλλά υπάρχουν πολλά άτομα τα οποία φεύγουν επειδή δεν υπάρχουν προοπτικές. Είναι άσχημες οι οικονομικές συνθήκες. Και ό,τι άποψη και να έχουμε, αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δικαιούνται άσυλο. Και εδώ πέρα έχουμε μια μεγάλη πρόκληση. Τι μπορούμε να κάνουμε για να στείλουμε πίσω αυτά τα άτομα με, και ακόμη περισσότερο με, για να είναι βιώσιμη η κατάσταση τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να μην προσπαθούν τα άτομα αυτά συνεχώς να μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ δεν έχουν πιθανότητες. Το ερώτημά μου λοιπόν προς την Κομισιόν είναι τι σκοπεύετε να κάνετε, τι κάνετε μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων, γιατί αναφέρθηκε ήδη ότι το να μιλάμε μόνο για αναπτυξιακή βοήθεια ή νόμιμες διόδους δεν θα είναι η λύση. Αλλά χρειαζόμαστε και άλλες απαντήσεις. Πώς λοιπόν γίνονται κάποιες συζητήσεις, π.χ. για να αλλάξει η γεωργική πολιτική, η εμπορική πολιτική, οι συμφωνίες ε, οικονομικής ε, εταιρικής σχέσης. Υπάρχει κάτι για να υπάρξει μία μόνιμη λύση και μία πραγματική συνεργασία με τις χώρες προέλευσης ή μιλάμε μόνο για τις ελάχιστες λύσεις που δεν ε, είναι μακροπρόθεσμες. Μάλιστα, Σοφή. Ευχαριστώ. Καλή χρονιά σε όλους. Μας γίνει το 2018 το έτος που επιτέλους θα έχουμε πραγματική, πραγματικό σύστημα αντιμετώπισης ε, και ανθρώπινο της μετανάστευσης. Για το θέμα που αναφέρθηκε βεβαίως το πραγματικό ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχει ε, το Συμβούλιο όταν μιλάμε για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν 28 κυβερνήσεις που πλακώνονται μεταξύ τους ε, με στόχο να είναι όσο δυνατόν πιο σκληρές και να το πασάρει μία στην άλλη. Ε, έχουν μάθει να παίζουν σε εθνικό επίπεδο και δεν ενδιαφέρονται ε, για να βρεθεί κάποια λύση. Γιατί νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές ότι μπορεί να γίνει. Ναι, μπορεί να γίνει. Αλλά βεβαίως είναι ευκολότερο να ασχολούνται ε, με τα θεωρία και τις κερκίδες. Αλλά πολλά έχουν ήδη ακουστεί. Πρώτα απ' όλα να ισχύσουν ε, τα όσα έχουν ε, νομοθετηθεί. Ναι, πράγματι. Αλλά θα πρέπει να ισχύσουν και οι φυστάμενοι κανόνες. Δεν μιλάω μόνο για την πολιτική ασύλου, αλλά και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, δεν χρειάζεται νομίζω να το πω. Τι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες κυβερνήσεις που δεν θεωρούν ότι δεσμεύονται από τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα όταν μιλάμε για τις πολιτικές ασύλου. Ε, κατόπιν νομίζω ότι θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο να μην φοβάται να επικοινωνήσει για τη μετανάστευση γιατί μπορούμε νομίζω να πούμε κάτι χωρίς συνεχώς να το λέμε ως, να το προσιάζουμε ως πρόβλημα. Δείτε τους φίλους μας στην άλλη όχθη εκεί, ε, του Ατλαντικού ε, οικονομήθηκαν από τη μετανάστευση. Εμεί γιατί υποθέτουμε ότι είναι πρόβλημα. Πρέπει να το διαχειριστούμε, ναι, να βρεθούν λύσεις, αλλά υπάρχουν και ιστορίες ε, επιτυχίας ε, και ωφέλους κτλ. Να τα λέμε και αυτά. Τα μιλήσατε για κατάχρηση του συστήματος και άλλοι το έθεσαν επίσης. Ναι, πράγματι χρειαζόμαστε νόμιμες διόδους. Ο κόσμος ο οποίος πάει σε άλλη χώρα για να βρει δουλειά δεν είναι εγκληματίας. Είναι έγκλημα να θέλει κανείς ε, καλύτερες συνθήκες ε, για την οικογένειά του. Ναι, ναι, βεβαίω πρέπει να διαχειριστούμε τη μετανάστευση, αλλά πρέπει να δώσουμε και τι ευκαιρίε. Και εμεί ω ε, κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε κάπως πιο επικριτικοί, γιατί χάνουμε και τις ευκαιρίες να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες. Και τέλος, συμφωνώ με την Τζιν Λάμπερτ. Όχι άλλες άτυπες και ανεπίσημες συμφωνίες, σας παρακαλώ. Και τέλος νομίζω ότι κάτι συμβαίνει, κάποιοι άνθρωποι σώζονται, αλλά ε, δεν ανέφερε κανείς ακόμα τα νησιά στην Ελλάδα. Έχουμε άτομα ε, τα οποία έχουν μετακινηθεί και έχουν φύγει από τα νησιά, αλλά χιλιάδες άνθρωποι έχουν κολλήσει εκεί σε άθλιες ε, συνθήκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καθαρά πολιτικούς λόγους. Για πολιτικούς λόγους. Δεν είναι ότι δεν είμαστε σε θέση να τους βγάλουμε από εκεί. Είναι για πολιτικούς λόγους. Λοιπόν, θα κάνουμε τα στραβά μάτια στην κατάσταση των ανθρώπων που ε, είναι εκεί πέρα, κρυώνουν, πεινάνε, έχουν πάθει κατάθλιψη και θα να αυτοκτονήσουν ή όχι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν μιλήσει ο Σάιμον και ο κύριος ε, Νίκολοφ, ε, να... να πω το εξής. Με το εξή. Οι συνάδελφοι είναι απεσιόδοξοι, γιατί βασίζονται βεβαίω στο ότι γίνεται στου τριμερεί διαλόγου και στη σκληρή δουλειά. Γιατί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση με το Συμβούλιο. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω η μπλε κάρτα από μόνη της δεν είναι ό,τι πιο σημαντικό. Αλλά αν δείτε αυτό το οποίο είπε η κυρία Κιέγγε για τις νόμιμες διόδους. Υπάρχει η εξής μία δηλαδή. Και οφείλουμε να επενέσουμε την Κομισιόν που έχει μια πολύ θετική στάση. Αλλά Εσεί ήσταν πολύ αισιόδοξο. Ε, πού βασίζεται αυτή η αισιοδοξία σας? Γιατί ε, με συγχωρείτε, δεν νομίζω ότι το κοινοβούλιο ε, θα μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο και να κάνει περισσότερες προσπάθειες όλες οι πολιτικές ομάδες. Δηλαδή, κάναμε ό,τι γινόταν αλλά αντιμετωπίζουμε, ας είμαστε ειλικρινείς. Τέλος εγώ είμαι πρόεδρος βεβαίως, δεν, δεν θα είμαι ειλικρινής. Θα σας παραπέμψω μόνο στα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Αυτά αντιμετωπίζουμε. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βλέπετε λοιπόν κάποια αισιοδοξία με βάση τα όσα βλέπουμε και από την Βουλγαρική Προεδρία. και κάτι άλλο για την μεταγκατάσταση. Ε, αναζητείτε κάποιο διαφορετικό αφήγημα, ε, χωρίς να διαφωνώ για τους αριθμούς. Αλλά εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι ε, τα κράτη-μέλη φταίνε. Μπορούμε να περάσουμε σε ένα αφήγημα που θα λέει ότι ε, ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους. Γιατί εγώ συμφωνώ με τα νούμερα τα οποία αναφέρατε αλλά ανησυχώ. Μάλιστα. Πολλές ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να απαντήσω. Θα απαντήσω σε όσες περισσότερες μπορώ. Η κυρία Κέγκε, τέλη Ιανουαρίου. Καλή υπενθύμηση. Ό,τι ζωή και να χαθεί στη Μεσόγειο είναι απώλεια. Είπατε στις 6 Ιανουαρίου 64 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Αλλά μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκή Ένωση στη διάσωση 620.000 ανθρώπων. Χάθηκαν φυσικά ζωέ, αλλά σώθηκαν και κάποιε και θα πρέπει να παραμένουμε σε παρύπνιση για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να εμποδίζουμε την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Και για την ερώτησή σας που συνδέεται με αυτή τη κυρίας Ιντφελτ για τα νομικά μα εργαλεία. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, διότι ακόμη τι αρμοδιότητες τι έχουν κυρίως τα κρατημέλη, είναι να συνδυάσουμε τις δυνάμεις των κρατών μελών και να τα φέρουμε αντιμέτωπα με τι ευθύνε τους τη πραγματικότητα. Αν εξηγήσουμε στους εταίρους μας ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να ε, εμποδίσουν τις παράνομες μετακινήσεις ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω νομιμοδών. Εάν δεν έχουμε απάντηση σε αυτό, πώς θα λάβουμε απάντηση στο επόμενο ερώτημα για τις νόμιμες οδούς ε, που προσπαθείτε να φτιάξετε. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε είναι αρκετά φιλόδοξο. Δεν ξέρω αν θα πετύχουμε, αλλά την ιδέα την ξεκινήσαμε από το Σεπτέμβρη. Να φέρουμε τα κάτι μέλη γύρω από το ίδιο τραπέζι και να πούμε ότι χρειάζεται με κάποιους από τους εταίρους μας, ε, με μια σειρά από χώρες, Βόρεια Αφρική λόγου χάρη, που ίσως εκεί υπάρχουν οι δυνατότητες στην αγορά εργασίας τους, που μπορούμε να συνδυάσουμε τις δικές μας δυνάμεις και έχουμε προηγμένες ε, μορφές συνεργασίας για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης, αλλά και χώρες νοτιούς της Σαχάρας. Σε αυτή τη φάση ενώ την Γκάμπια, ας πούμε, ή την Γουινέα ή τον Ιγυρά να δούμε ε, τι ε, αξιο... τι ε, δυνατότητες μπορούμε να αξιοποιήσουμε από τη δική τους χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να καλύψουμε την ε, ζήτηση που υπάρχει δημιουργώντας νόμιμες οδούς για την ε, υποδοχή μεταναστών σε συγκεκριμένους τομείς που μπορεί να τους χρειαζόμαστε. Αυτές τις συζητήσεις κάνουμε με τα κρατη προσπαθώντας την... την μπορούμε να πετύχουμε στη συνεργασία μεταξύ τους και πώς τους επόμενους μήνες ως το Μάιο μπορούμε να ξεκινήσει ένα τέτοιο εγχείρημα. Αυτό που μπορώ λοιπόν να κάνω είναι να δεσμευτώ εγώ ή οι συνάδελφοι που εργαζόμαστε επί του θέματος να ξαναέρθουμε να σας κάνουμε μια παρουσίαση για το πώς προχωράμε στο θέμα αυτό, τι βήματα έχουμε κάνει στη σχετική πορεία. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η χρηματοδότηση, τα κονδύλια στο συνδυασμό των δυνάμεων των κρατών μελών. Διότι κάτι το περίεργο στο όπω και να το κοιτάξει κανεί αυτό, είναι ότι πολλά γίνονται σε εθνικό επίπεδο, αλλά σπανίω συνδυάζονται με τρόπο συνεπή και συνεκτικό. Ε, χρειάζεται λοιπόν να ε, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη επιρροή και επίδραση με τις προσπάθειε που ούτω ή άλλω γίνονται, να γίνονται με τρόπο κοινό. Αυτά αναφέρονται και στο έγγραφο και θα μπορούσα να σα δώσω περισσότερα στοιχεία εκτό εφόσον θέλετε και σα ενδιαφέρει. Ε, έχουμε ε, συμφωνία για το μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό, τον οργανισμό, πέρυσι το καλοκαίρι. Οπότε ε, περιμένουμε μέχρι το Μάρτιο να υιοθετηθεί, γιατί και εδώ έρχομαι στην απάντηση προς την κυρία Λάμπερτ. Αυτό θα επιτρέψει και στον οργανισμό να αρχίσει να ενισχύεται, να δυναμώνεται, να συγκροτηθεί και να ετοιμαστεί, ώστε όταν ε, υιοθετηθεί και μεταρρυθμίσει του συστήματος του Δουβλίνου να ξεκινήσει αμέσω. Και επανέρχομαι και στο ζήτημα τη κυρία ε, Ιντβέλτ. Όσο εκκρεμεί το Δουβλίνο θα έχει ο οργανισμό ε, διευρυμένη δυνατότητα παρακολούθηση. Αυτό προβλέπει και το καταστατικό. όσο εκκρεμεί η συμφωνία αυτή, θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά αυτό που προβλέπει τη δύστη νομοθεσία, κάτι που δεν ισχύει πάντα. Πίτερ Νίτερ Μίλλερ, διαφωνώ σε ένα θέμα μαζί σου όπως είπαν και ο Κλώτ και η ίσως θα ήταν άδικο να κατηγορούμε μόνο την Εστονική Προεδρία, γιατί έκαναν πραγματικές προσπάθειες και κόπιασαν ε, στην Προεδρία, αλλά δεν υπήρχε η απαραίτητη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη για να σημειωθεί πρόοδος. Δεν φταίει γι' αυτό η Εστονική Προεδρία και ίσως η αισιοδοξία μου οφείλεται και στο ότι μόλις τώρα γυρίζω από τι χριστουγεννιάτικε διακοπέ, Πάντως πιστεύω ότι υπάρχει σε επίπεδο ηγετών αποφασιστικότητα και βούληση να υιοθετηθεί η μεταρρυθμίση του Δουβλίνου και ένα κοινό σύστημα ασύλου για να έχουμε ένα, μια μακροπρόθεσμη, διαχειρίσιμη και βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που δεν θα στηρίζεται σε μεμονωμένες αποφάσεις που δεν θα είναι και πολιτικά βιώσιμες. Γι' αυτό πιστεύω ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία και με το πρόγραμμα των ηγετών αλλά και με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μίλησε για πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Κορυφής του Ιουνίου. Είναι όλα καλά, αλλά φυσικά χρειάζεται περαιτέρω έργο γιατί ό,τι ε, συμφωνία και προκύψει του συμβούλιο. θα διαφέρει σημαντικά σε πολλούς τομείς από τη δική σας θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει λοιπόν να επιτύχουμε στη συνέχεια μία συμφιλίωση των δύο απόψεων, κάτι που προϊονίζει δύσκολες ερωτήσεις. Κυρία Σπινέλη, δεν ήθελα να δώσω την εντύπωση ότι η μείωση του αριθμού των παράτυπων αφήξεων, η αύξηση της Επιτροπής των Επιστροφών είναι μία ανθρωπιστική ε, πρόοδος, ανθρωπιστικό επίτευγμα. Απλώς αποτελεί ένα ε, ένα τμήμα τη φερική μας προσέγγιση για τη μετανάστευση, ώστε όσοι χρήζουν προστασία να λάβουν τέτοια προστασία και ιδεοδός μέσω τη επανεγκατάστασης και όχι πληρώνοντα ένα διακινητή για την ε, παράνομη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να πω. Είναι τμήμα της φερική μα προσέγγιση. και θα ήθελα να διατρανώσω ότι δεν γίνεται καμία επιστροφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Λιβύη. Το διαψεύδω αυτό κατηγορηματικά ότι υπάρχουν τέτοιες επιστροφές. Συνεργαζόμαστε με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και με, το, την Ορμοσία των Προσφύγων ώστε να έχουμε ε, οικειοθελείς επιστροφές σε ένα συνολικό αξιοπρεπές πακέτο. Και όσοι θέλουν ε, εκούσια κάποιοι να επιστρέψουν στη Λιβύη και φυσικά δεν ζητούν προστασία ή άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για τους ετούντες άσυλο και πάλι ε, συνεργαζόμαστε με τους οργανισμούς του ΙΕ και μάλιστα είχαμε κατεπίγουσα εκένωση ε, ανθρώπων από τη Λιβύη προς τον Ήγυρα και μετά από τον Ήγυρα ε, για επανεγκατάσταση με καθεστώς προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένας όμως δεν έχει επιστραφεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ τη Λιβύη. Για τον Νίγηρα δεν ξέρω τι κάνουν και τα κράτη-μέλη, στρατιωτικέ επιχειρήσει. Αυτό μπορώ να σα πω είναι ότι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συνεργάζεται με τις αρχές του Νίγηρα για να ενισχύσουμε τι δραστηριότητε, τις ικανότητές τους να εξαρθρώσουν κάποια κυκλώματα διακινητών ή σωματεμπόρων Επίσης, προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες κοινωνικές και οικονομικές εναλλακτικές προς, το, προς την λαθροδιακίνηση σε περιοχές όπως τα Κατές και συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές του Νίγηρα για την προστασία των συνόρων. Επίσης, έχει μειωθεί ο αριθμός αφήξεων από, τη, από το Νίγηρα στη Λιβύη και έχει μειωθεί από 70.000 σε 7.000 το μήνα ο αριθμός αυτός. Τώρα έρχομαι στην ερώτηση της κυρίας Μετσόλα που ε, απήχησε κάποια σημεία των, κυριών Σίπελ και ε, Ιντφελτ. Ένα από τα θέματα αυτά ήταν η εφαρμογή του σχεδίου εξωτερικών επενδύσεων για την κινητοποίηση 44 δισεκατομμυρίων ευρώ ιδιωτικών επενδύσεων, κυρίως στην Αφρική και θα δημιουργήσουν νομίζω σημαντικές ευκαιρίες εργασίας και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει για να σημειωθεί η πρόοδος σύντομα. Κυρία Γκραπίνη, αν είναι όλα τέλεια, όχι, όχι, όχι βεβαίω. μακράν αυτού. Να σας δώσω δύο παραδείγματα. Αν δείτε παραδείγματος χάρη το ποσοστό αναγνώρισης για Αφγανούς κυμαίνεται από 99% μέχρι 0%. Εν δηλαδή, Υποτίθεται ότι έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι το ίδιο το νούμερο παντού, αλλά δεν υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των δύο αυτών αριθμών. Και επίσης ε, βλέπουμε ότι οι διαδικασίες ε, κρατάνε από λίγους μήνες περιλαμβανομένης ε, και της προσφυγής μέχρι χρόνια σε κάποια κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε μέσω του κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου και των εκθέσεων αυτών. Αλλιώς ε, υπάρχει ένα κίνητρο να επιλέγει κάποιος που θα υποβάλει αίτηση για άσυλο. Για την ερώτησή σας για τις προσδοκίες μου για την δήλωση με την Τουρκία θα περιοριστώ στην πτυχή της μετανάστευσης. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξο ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί η δήλωση αυτή και ότι δεν θα δούμε τεράστια αύξηση των αφήξεων. Ε, κυρία Λάμπερτ, εάν ε, είναι σωστός ο προπολογισμό για την ΕΑΖΟ σε σύγκριση με την συνοριοφυλακή, πρώτα απ' όλα θα έλεγα ότι η Frontex ήδη έχει μεταβληθεί στην υπηρεσία αυτή με επιπλέον ε, αρμοδιότητες. Τώρα δεν ξέρω αν έχει λυθεί το πρόβλημα στο Συμβούλιο με την υπηρεσία ασύλου αυτό θα απαιτήσει περισσότερα κονδύλια ακόμα για την υπηρεσία συλλογή, γιατί υπάρχουν νέα καθήκοντα και νέες ευθύνες. Υπάρχει ένας ενισχυμένος ρόλος επιτήρησης, στήριξης και ταυτόχρονα βεβαίως το ίδιο βλέπουμε και στην υπηρεσία στην φυλακής. Θα έλεγα όμως το εξής ότι όσο δεν υπάρχει ακόμα η υπηρεσία και όσο τα κράτη-μέλη δεν προσφέρουν πάντα την στήριξη που χρειάζεται η Ελλάδα και η Ιταλία θα πρέπει να χρηματοδοτεί η ΕΑΖΟ για να δίνει μια στήριξη πρώτης γραμμής σε Ιταλία και Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι το Κοινοβούλιο έχει ένα ρόλο στην εφαρμογή της δήλωσης με την ε, Τουρκία και βεβαίως ε, κάτι πρέπει να γίνει και για το θέμα αυτό της διαχείρισης των 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και υπάρχει βεβαίως και το θέμα της απελευθέρωσης της βίζας ε, οπωσδήποτε θα γίνει σεβαστός ο ρόλος του Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση των επιστροφών και το τι συμβαίνει κατόπιν τα περισσότερα από αυτά γίνονται στο πλαίσιο μιας σύμβαση με τον Διεθνή Οργανισμό μετανάστευση και η υποχρέωσή τους είναι ακριβώς η παρακολούθηση του τι συμβαίνει μετά. Γιατί βεβαίω υπάρχουν, ε, αυτό το οποίο είπε και η κυρία Λάμπερτς, διαφορετικέ προσδοκίες για το τι θα συναντήσει ο κόσμο που επιστρέφει στη Λιβύη σε σχέση με το τι βρίσκει εκεί. Κυρία Σίπελ, έχετε δίκιο. Ε, είπατε και εσείς και η κυρία Ινετφέλντ έχουμε δύο επιλογές. Μπορούμε να δούμε τη μετανάστευση ως απειλή ή ως ευκαιρία. Η μετανάστευση δεν θα εξαφανιστεί. υπάρχει, υπάρχει και η υποχρέωσή μας νομίζω να το θεωρήσουμε ευκαιρία και να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τη μεταναστεύση. Αυτό περιλαμβάνει και την αναπτυξιακή βοήθεια και μια ανάπτυξη νομίζω του εξωτερικού ταμείου επενδύσεων και νόμιμες διόδους και βεβαίως οργανωμένες νόμιμες διόδους για όσους θέλουν να εργαστούν και να ζήσουν και οι ίδιοι καλύτερα. Πρέπει νομίζω επίσης να δούμε το τι γίνεται με τις εμπορικές μας σχέσεις. Έχουμε κάνει αρκετά πράγματα και νομίζω ότι έχει σημειωθεί επίσης πρόοδος και στην γεωργική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι κάτι το οποίο γνωρίζω ότι εξετάζει η Επιτροπή Ανάπτυξης και συμφωνώ πλήρως. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια ολιστική προσέγγιση με τους Αφρικανούς εταίρους μας. Για την ερώτηση της κυρίας Ινετφέλντ για το τι κάνουμε για την εφαρμογή των κανόνων που υπάρχουν ήδη κάτι το οποίο δεν απασχολεί τον τύπο. Την ίδια ημέρα που εγκρίναμε αυτήν την ανακοίνωση. όχι το πρώτο βεβαίως απασχόλησε τον τύπο, Πολωνία, Τσεχία, ε, προσφύγαμε στο δικαστήριο κατά αυτών των χωρών ε, για την υποχρέωσή τους για την μεταγκατάσταση, και ε, με την Ουγγαρία συνέβη το ίδιο για το σύστημα ασύλου και την ζώνη διέλευσης που σαφώς δεν συμφωνεί με το κεκτημένο. Και είναι υποχρέωσή μα ω θεματοφύλακα τη συνθήκη. Και έχουμε και κάποιε άλλε διαδικασίε ε, που είναι ανοιχτέ και έχουμε παρομοίε ανησυχίε με άλλα κράτη-μέλη, κάτι το οποίο βεβαίω παίρνουμε πολύ σοβαρά. Το να μην υπάρχει συμφωνία για το διπλίδωνο δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να μην εφαρμόζει την υφιστάμενη νομοθεσία για τα ελληνικά νησιά. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Συνεργαζόμαστε με τις ελληνικές αρχές τους τελευταίους μήνες. Δώσαμε πολύ σημαντική οικονομική στήριξη 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ στις ελληνικές αρχές. Ε, καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες. Να σας δώσω ένα πρακτικό παράδειγμα. Ε, ο κόσμος στα νησιά φεύγει από τα στρατόπεδα και πάει σε νοικιαζόμενα ε, σπίτια, τα ξενοδοχεία έχουν γεμίσει. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να γίνει κατεπηγόντως είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει κόσμο στην Τουρκία όταν απορρίπτεται η αίτηση ασύλου, κάτι το οποίο δεν κάνει αυτή τη στιγμή για διάφορους λόγους. Νομίζω ότι έτσι θα μειωθεί πολύ η πίεση στα νησιά. Τέλος, για τις ε, ερωτήσεις του Πρόεδρου. Μπλε κάρτα, αισιοδοξία. Η αισιοδοξία μου πηγάζει από το ότι αναγνωρίζω αναγνωρίζουν τα κράτη-μέλη ότι το να μην υπάρχει κανένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα δεν μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται ως κατάσταση. Ελπίζουμε έτσι να υπάρξει κάποια αλλαγή και να υπάρξει μπλε κάρτα, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουν και τα κράτη-μέλη ότι χρειάζεται περισσότερη Ευρώπη σε κάποιους από αυτούς τους τομείς, γιατί Χωρίς αυτό πολύ δύσκολα θα επιτύχουμε συμφωνία σε αυτά τα ζητήματα γιατί δικαίως λέτε ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη εναρμόνιση ε, στα ζητήματα αυτά. Τέλος, για την ε, μετακαταστάση. Ε, η αριθμή είναι χαμηλή, γεγονός, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια επιτυχής εφαρμογή των ατόμων που είναι επιλέξιμο για αλλά υπάρχουν προβλήματα. Εγώ δεν είμαι υπέρ του κατοφλίου 75%. Πρέπει να διορθωθεί αυτό στο Δουμπλίνο και η Ελλάδα και η Ιταλία χρειάζονται άλλη αλληλεγγύη και σήμερα. Και τα κράτη-μέλη κάνουν πάρα πολύ δουλειά προ όφελο των 28 και πρέπει να γνωρίζουν ότι αν υπάρξει κάποια στήριξη θα έχουν στήριξη. Αν υπάρξει κάποια κρίση θα έχουν τη στήριξη μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Νίκολοφ ε, συμφώνησε να μην μιλήσει γιατί βεβαίω έχουμε καθυστερήσει. Και έχουμε, και, έχουμε και προσκεκλημένους που περιμένουν να λάβουν το λόγο. Δεσμότατε Μπάντιο αν θέλετε να έρθετε στο Προεδρείο. Και εσείς συνάδελφοι μείνετε στην αίθουσα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μόντιου. Συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη από τους προσκεκλημένους μας που ξεκινάμε τόσο αργά το σημείο αυτό που είναι τόσο σχετικό, αλλά σας παρακαλώ εσάς να μείνετε και θα αρχίσω να κάνω την εισαγωγή μου όσο κάθονται οι προσκεκλημένοι μας. Απόκριση στα 20 σημεία δράσεις για το Παγκόσμιο Σύμφωνο απόκριση στα ζητήματα των προσφύγων και των μεταναστών. Όλα αυτά ξεκίνησαν με συζητήσεις πριν από την σύνοδο του Port Francis, την πρώτη δήλωση δηλαδή του Κοινοβουλίου τον Έμβριο. και είμαστε σε συνεννόηση με την Αγία Έντρα, ε, και μετά την πρώτη δήλωση του Παπαφραγκίσκου Ο τίτλος του θέματος αυτού είναι ε, το έγγραφο του Τμήματος Μεταναστών και Προσφύγων της Αγίας Έδρας για το θέμα των προσφύγων και μεταναστών. Και θέλαμε να μας παρουσιάσει ο αδερφός Μπάντζιο την, ε, τα όσα έχει να μας πει σε σχέση με το θέμα αυτό και την απόκριση για τα ζητήματα προσφύγων και μεταναστών. Έχετε το λόγο. Να ξεκινήσω ευχαριστώντας για την ε, ευγενική πρόσκληση που έλαβα. Και εδώ ήθελα να παρουσιάσω αυτά τα 20 σημεία δράσης για το θέμα των μεταναστών και των προσφύγων που ετοίμασε η δική μας υπηρεσία ως συνεισφορά για την όλη διαδικασία που θα μας ε, οδηγήσει προς την υλοποίηση του συμφώνου το 2018. Έχω ετοιμάσει και μια σειρά από διαφάνειες για να μας βοηθήσουν. Με την επιστολή του και το κείμενο «Manam Progressionem» για την ανθρώπινη πρόοδο, ο Πάπας Φραγκίσκος ε, εξέφρασε τις σχετικές του απόψεις. περνώντας από την μετακίνηση των ανθρώπων στις υγειονομικές τους ανάγκες. Ε, υποστηρίζει ότι χρειάζονται εργαλεία ε, βιώσιμη ανάπτυξη για την ε, προστασία των ανθρώπων αυτών και με τις κρίσεις κρίσει που νομοτοπίζουμε τα τελευταία χρόνια λόγω της πίεσης της αύξηση του πληθυσμού, των, των φυσικών καταστροφών και τη προσοχή που πρέπει να δώσουμε πλέον στη μετακίνηση των μεταναστών και προσφύγων. Γι' αυτό η ιδιαίτερη μνήμα στα ζητήματα προσφύγων και μεταναστών. Στην υπηρεσία αυτή άλλωστε την ε, γίδα έχει ο ίδιος ο Πάπας και η Εκκλησία σκοπό έχει να λειτουργήσει υπό την αιγίδα του ε, Αγίου Πατέρα ως ε, οδηγός στα θέματα αυτά. Η υπηρεσία για τους μετανάστευσης και τους πρόσφυγες ε, κάνει ξεκάθαρη μια από τις βασικές αποστολές της Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή να συνεδρεί τους ανθρώπους σε όλες τις στιγμές της ζωής τους, είτε είναι οδύνης, χαράς, ε, αγωνίας, άγχους τους και αυτούς που υποφέρουν. Μεγαλύτερη αποστολή της υπηρεσίας είναι να στηρίζει την Εκκλησία σε τοπικό επίπεδο, διεθνές ε, και τοπικό, για να παρακολουθεί την μεταναστευτική πορεία όλων αυτών των ανθρώπων με ιδιαίτερη προσοχή όσων για διαφορετικούς λόγους αναγκάζονται να μετακινηθούν ή να διαφύγουν. Αυτή καθεαυτή η Καθολική Εκκλησία έχει δώσει βοήθεια με ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα τα οποία μπλέκονται σε αυτέ τι ανθρωπιστικέ δραστηριότητε. Σήμερα, ενώ έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων ανθρώπων και μεταναστών προσφύγων στην σύγχρονη ιστορία, η Καθολική Εκκλησία συνεχίζει να διευθύνει αυτό το έργο σε ε, αλληλεγγύη με του εκτοπισμένου, μετακινούμενου και τη διεθνή κοινότητα. Ενώ τεράστιε μάζε ανθρώπων αναγκάζονται να αφήνουν τι αιστείε του και τι οικογένειέ του λόγω διωγμών, βία, φυσικών καταστροφών και τη μάστιγα τη φτώχεια. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η μετανάστευση είναι μια φυσική ανθρώπινη αντίδραση σε κρίσεις και είναι και μία απόδειξη ότι υπάρχει ε, έμφυτη ανθρώπινη επιθυμία να αναζητά κανείς την ευτυχία και να απολαμβάνει μια καλύτερη ζωή. Η πραγματικότητα αυτή έχει σημαντικότητα τι πνευματικέ και οι προεκτάσει. και υπάρχει σοβαρό αντίκτυπο στι συμπεριφορέ και τι αντιδράσει των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και στην τωρινή κρίση οι εμπειρίε μα μας δείχνουν ότι μπορούμε να βρούμε κοινέ αποκρίσεις και αποτελεσματικέ και η Εκκλησία σκοπό έχει να συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για να προωθήσει και να υιοθετήσει δραστικά μέτρα ε, πρόθεση τη αξιοπρέπεια, τη σεβασμού των δικαιωμάτων και τη ελευθερία, όλων των όσων συμμετέχουν στις μετακινήσεις αυτέ πληθυσμών, εκτοπισμένων, εσωτερικώς εκτοπισμένων μεταναστών και προσφύγων οι διαδικασίες που έχουν ξεκινήσει από τον ΟΗΕ για την εκπόνηση του διεθνούς Παγκόσμιου Συμφώνου με ιδιαίτερη στου ε, πρόσφυγε και μετανάστε είναι μια μοναδική ευκαιρία για να δώσουμε μια κοινή απάντηση ω προ τη διεθνή συνεργασία και τι κοινέ ευθύνε που όλοι πρέπει να αναλάβουμε. Η Εκκλησία έχει εκφράσει επανειλημμένω το δικό τη ενδιαφέρον για του όρου που θέλουμε να περιλαμβάνει το Παγκόσμιο Σύμφωνο και βάσει τη μακροσκελού τη εμπειρία μπορεί να δώσει πολλέ χρήσιμε συνεισφορέ σε αυτή την διαδικασία. Το Βατικανό με διάφορες επισκοπικές ε, συγκλήτους, ε, συνόδους μάλλον για το θέμα αυτό, έχει εκπονήσει τα 20 σημεία που θα σας παρουσιάσω εδώ, που έχει εγκρίνει Άγιος Πατέρας, που βασίζονται σε καλές πρακτικές ως τώρα και που είναι μια χειροπιαστή απόκριση της Καθολικής Εκκλησίας στις ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών και που σκοπό δεν έχουν να εξαντλήσουν την προσφορά της Εκκλησίας για τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης, αλλά είναι μια σειρά από πρακτικές συμβουλές που όσοι δρούν στα πλαίσια της Καθολικής Εκκλησίας δεν μπορούν παρά να χρησιμοποιήσουν και να συμπληρώσουν στο έργο τους και στον καθημερινό τους διάλογο με τις κυβερνήσεις ε, στην φάση της υλοποίησης του Παγκόσμιου Συμφώνου. Τα 20 σημεία σημειώνουν μια σειρά από αποτελεσματικές ιδέες που σκοπό έχουν να δώσουν μια ενιαία απάντηση στις σημερινές προκλήσεις σε συνεργασία με ε, ε, τον Πάπα Φραγκίσκο. Ο σκοπός είναι να προστατευθούν, να ενσωματωθούν, να προαχθούν και να ενταχθούν οι πρόσφυγες. Ξεκινάμε από όσα είναι εφικτά σε αυτή τη φάση για να περάσουμε στον τελικό σκοπό, δηλαδή να δημιουργηθεί ένα κοινό οίκο στον οποίο μπορούν να ζουν και να ευημερούν όλοι. Η ελπίδα μα είναι ότι όσα προτείνονται θα είναι ε, ένα γνώμονα για όλου του πολιτικού ηθήνοντε και για όσου ασχολούνται με τα θέματα προσφύγων και μεταναστών, ετούντε άσυλο και εσωτερικώ εκτοπισμένων και κυρίω για του πιο ευάλωτου. Τα ε, στοιχεία δείχνουν ότι η μετανάστευση όλο και περισσότερο αποτελείται από ροέ μεικτέ. Είναι δύσκολο να κάνει κανεί μια σαφή διάκριση μεταξύ μεταναστών και προσφύγων. Διότι πολλέ φορέ τα κινητρά του για τη μετακίνηση είναι παρόμοια αν όχι επανομοιότυπα. Οπότε ο σκοπό είναι να δούμε του όρου διαπραγμάτευση και ε, ε υλοποίηση του Παγκόσμιου Συμφώνου, γιατί ο σκοπό είναι να κάνουμε μια πραγματική διαφορά για τι ζωέ των ανθρώπων αυτών, με μεθόδου και σκοπού που θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω μηχανισμών αξιολόγηση και των αποτελεσμάτων. Το τμήμα των μεταναστών και προσφύγων της Αγίας Έντρας έχει σκοπό να ε, προωθήσει την ε, υλοποίηση των 20 σημείων στο τέλο του 2018 με την Προεδρία του Παπαθαγίσκου για την ενίσχυση τη διεθνού κοινότητα, Ελπίζουμε τα 27 σημεία να συμπεριληφθούν και ρητό στο Παγκόσμιο Σύμφωνο. Τα ίδια τώρα τα σημεία δράση και να πω απλώ ω υποσημείωση ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση στι προπαρασκευαστικέ ε, συνεδριάσει του Παγκόσμιου Συμφώνου συνεισέφερε ε, σημαντικά στην ε, σύνταξη του εγγράφου. Θα δείτε κι εσεί από μόνοι σα διαβάζοντα το έγγραφο που υπάρχουν συμπτώσει απόψεων. Υποδοχή ανάπτυξη των νόμιμων και ασφαλών οδών για του νόμιμου μετανάστε. Η απόφαση τη μετανάστευση είναι ελεύθερη και οικειοθελή. Θα πρέπει η μετανάστευση να γίνεται με το σεβασμό τη κάθε ενδιαφερόμενη χώρα, με το σεβασμό τη νομοθεσία τη κάθε ενδιαφερόμενη χώρα. Η Εκκλησία προτείνει τα εξή, να μην υπάρχει ομαδική απέλαση προσφύγων και μεταναστών που ε, δεν βασίζεται στον νόμο. Πάντοτε να γίνεται σεβαστή η αρχή τη μη ε, επιστροφή σε χώρε που δεν θεωρούνται ασφαλεί. Η αρχή αυτή βασίζεται στην ασφάλεια που μπορεί πραγματικά να προσφερθεί στο άτομο και όχι σε μια συγκυριακή αξιολόγηση της γενικής ασφάλειας της χώρας. Δύο. Παροτριούνται τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις νόμιμες οδούς για μια ελεύθερη και οικειοθελή μετανάστευση, όπως και ο, ε, η μετακατάσταση των προσφύγων πρέπει να γίνεται με θεωρήσεις για μετανάστες φοιτητές, ερευνητές και φοιτητές. Για τους φτωχούς και πλέον ευάλωτους, για την... Ε, υλοποίηση προγραμμάτων για την ένταξη των προσφύγων, την προσφορά θεωρήσεων για, τον οικογενειακό, ε, για την οικογενειακή επανένωση με ε, γονείς, παππούδες και θείους ή με, τις ιδιαίτερη, με την ιδιαίτερη μέρημνα για όσους ε, προσπαθούν να ξεφύγουν από περιοχές με εχθροπραξίες, πολεμικές συγκρούσεις ή τις όμορες, τις μεθοριακές περιοχές. Θα πρέπει εδώ να λαμβάνεται υπόψη σε κάθε περίπτωση η προσωπική ασφάλεια των ατόμων και όλων των ετούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στην επικράτεια μιας χώρας. Αυτό μπορεί να γίνει με την απαραίτητη εκπαίδευση των συνοροφυλάκων, και τις ε, εγγυήσει πρόσβασης όλων των μεταναστών, των άσυλο και προσφύγων με όρους ε, προστασίας για όσους αποδρούν από περιοχές με ε, πόλεμο ή συγκρούσεις και φτάνουν στην εθνική επικράτεια ενός κάτω μέλους χωρίς να έχουν τη σχετική έγκριση. Επίση, θα πρέπει να προασπιζόμαστε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των προσφύγων και μεταναστών. Η Εκκλησία υπογραμμίζει την ανάγκη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ολιστική όπω ονομάστηκε σε προηγούμενε συζητήσει, για τα θέματα τη μετανάστευση. Θα πρέπει στο κέντρο να βρίσκεται το ε, ανθρώπινο όν ε, με σεβασμό τη αξιοπρέπεια και των δικαιωμάτων. Το δικαίωμα στη ζωή είναι το πλέον βασικό και χωρί την άσκηση αυτού του δικαιώματο δεν ε, μπορεί να. Μάλλον η άσκηση του δικαιώματο αυτού δεν μπορεί να εξαρτάται από το καθεστώ του καθεστώς ενός ανθρώπου προς τη μετανάστευση. Οι αρχές των χωρών προέλευσης καλούνται να προστατεύσουν τους πρόσφυγές τους με την προσφορά ε, τεκμηριωμένων πληροφοριών πριν την αναχώρηση. Θα πρέπει επίσης να οργανωθούν ανάλογοι οργανωσμοί μετανάστευσης με την εμπλοκή του αρμόδιου Υπουργείου που ασχολείται με τα θέματα ε, μετανάστευσης και την ε, συμμετοχή του Υπουργού του Υπουργείου Εξωτερικών. Επίση, οι χώρε αύξηση θα πρέπει να προστατεύουν τι πρόσφυγε για να εμποδίσουν την εκμετάλλευσή του και την. Ε, και με την ε, απέτηση προς τους εργοδότες να ζητούν ε, νόμιμα στοιχεία ταυτοποίησης των μεταναστών ασχέτως με το καθεστώς τους και χωρίς αρνητικές συνέπειες για την περαιτέρω διαμονή τους. Η δυνατότητα να ανοίξουν προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και να πληρώνονται τουλάχιστον μία φορά το μήνα είναι απαραίτητε συνθήκε. Καλούνται τα κρατημέλη, αριθμό 6, να ζητήσουν από του μετανάστε και του ετούντε άσυλο αλλά και του πρόσφυγε συνθήκε ώστε να μπορούν να ασκήσουν καλύτερα τι ε, δεξιότητέ του και να αξιοποιήσουν τα προσόντα του προ όφελο τη τοπική κοινότητα. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τη εγγύηση τη ελευθερία κυκλοφορία εντό μια χώρα, την προσφορά άδεια εργασία, την συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στην υποδοχή των των άσυλο, την πρόσβαση σε μέσα επικοινωνία και την ανάπτυξη προγραμμάτων επανένταξη κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα για όσου αποφασίσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα του. Έβδομο, τα κράτη-μέλη καλούνται να προστατεύσουν του ανήλικου που είναι πλέον ευάλωτοι, του μείον τους, τους ε, συνόδευτους μάλλον ανήλικους και όσους δεν συνοδεύονται από μέλη της οικογένειάς τους βάσει του δικαίου, του παγκόσμιου δικαίου για τα παιδιά. Αυτό πρέπει να γίνει με τον εντοπισμό εναλλακτικών λύσεων προ την κράτηση των ανηλικών μεταναστών που βρίσκονται σε συνθήκε παρανομία. Θα πρέπει να προβλεφθεί μια προσωρινή κυδαιμονία ή κάποιο είδου προστασία για του ανήλικου που είναι ασυνόδευτοι ε, ή μόνοι και ε, να βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ενηλίκων ε, ή θα πρέπει επίσης βάσει της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών να ε, προστατευθούν οι ανήλικοι που δεν θα πρέπει να κηρύσσονται παράνομοι πριν την ε, έλευσή τους στην ε, ηλικία της ενηλικίωσης. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη να προσφέρουν ε, εκπαίδευση, πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλου του ανηλικού πρόσφυγε μετανάστε και του άσυλο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, ασχέτω του καθεστώτος του μετανάστευση με τρόπο ίδιο προ του ε, ηθαγενεί πολίτες μιας χώρας. Επίσης καλούνται τα κράτη να προσφέρουν στου πρόσφυγε και μετανάστε, πρόσβαση στο κράτο ε, πρόνοια με την ε, υγειονομική περίθαλψη ε, που αναλογεί και στους πολίτες μιας χώρας. Ακόμη και πρόσβαση στα συνταξιδοτικά συστήματα μιας χώρας και ε, την προσφορά των ανάλογων δικαιωμάτων εφόσον επαναπατριστούν. Θα πρέπει να αποφύγουμε να είναι απάτριδες οι πρόσφυγες και μετανάστες βάσει των διεθνών συμβάσεων και να τους δοθεί ηθαγένεια, ιδίω στα παιδιά, τη στιγμή της γέννησής τους. Βάσει και της δήλωσης για τα δικαιώματα των νηπίων. Εδώ θα πρέπει να ευνοηθεί η ανθρώπινη εξέλιξη των μεταναστών και προσφύγων. Η Εκκλησία εντοπίζει την ανάγκη να προσθεθεί ή να ε, καλλιεργηθεί η ολοκληρωμένη ανθρώπινη πρόοδο των μεταναστών και προσφύγων, όπω και στο υπόλοιπα μέλη μια τοπική κοινότητα. Σε όλε τι χώρε, οι έντοντε άσυλο πρόσφυγε και μετανάστε πρέπει να έχουν πρόσβαση στο ε, κράτο, ε, και στις δομές του και καλούνται τα κράτη να γνωρίσουν και να δώσουν στους πρόσφυγες σε άσυλο και μετανάστες τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους στο κράτος άφηξής τους. Μέσω των, της πρόσβασής τους στο εκπαιδευτικό σύστημα ή περαιτέρω προγραμμάτων, ε, στάζ και άλλων ασκήσεων και μαθητιών, όπως ισχύουν στα οικία κράτη, και βάσει των τίτλων σπουδών που έχω αποκομίσει αλλού. Επίσης τα κατημέλη καλούνται να επιτρέψουν την εργασιακή και κοινωνική ένταξη των ετούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών στις τοπικές κοινότητες μέσω της αναγνώρισης της ελευθερίας κυκλοφορίας τους και επιλογής του τόπου διαμονής τους. Θα πρέπει να τους δοθεί δυνατότητα να εργάζονται και σε όλους να προσφέρονται, όπως και τα μέλη της τοπικής κοινότητας, η πρόσβαση ε, ε, στην ζωή της τοπικής κοινότητας και πληροφορίες στην ε, μητρική τους γλώσσα. 14. Τα κράτη-μέλη καλούνται να προστατεύουν την αξιοπρέπεια και την ενότητα των οικογενειών, ασχέτω ε, του καθεστώτο του ω προ μετανάστευση. Αυτό επιτρόποντας την διευρυμένη επανένωση των οικογενειών και βάσει των οικονομικών απαιτήσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας της επανένωση να εργάζονται και, ε, και επανενώνοντα ε, μέλη της οικογένειας που έχουν βρεθεί σε διαφορετικέ χώρε. Θα πρέπει οι ανήλικοι να προστατεύονται και βεβαίω η οποιαδήποτε εργασία των μελών της οικογένειας να μην είναι εις βάρος της υγείας και της εκπαίδευσης των ανηλίκων. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικέ ανάγκες και το ευάλωτο των ε, ανθρώπων αυτών και να δίδονται τα δικαιώματα του πολίτη κανονικά και με βάση τις ειδικέ του ανάγκες εφόσον είναι ανάπηροι ή έχουν ειδικέ ανάγκες. Είτε είναι ενήλικοι είτε ανήλικοι και με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα όπως και για τους ε, πολίτες μιας χώρας. Θα πρέπει η διεθνή συνεργασία να ενταθεί στο επίπεδο της ανθρωπιστικής συνεργασίας και οι χώρες που δέχονται μεγάλες ροές προσφύγων και μεταναστών να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να μπορούν όλοι να υποφεληθούν ασχέτως του καθεστώτο αυτός ως πρώτη μετανάστευση. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρηματοδότηση δομών, υποδομών, ιατρικής περίθαλψης, κοινωνικής στήριξης και ένταξης στις χώρες άφηξης που θα πρέπει να προσφερθούν στους ενδιαφερόμενους και στις τοπικές κοινότητες. Επίσης, καλούνται τα κράτη να εξασφαλίσουν την άνεξη θρησκεία θεωρητική και πρακτική σε όλους τους ετούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστευσης, ασχέτως με το καθεστώς τους ως προς τη μετανάστευση επανένταξη. Θα πρέπει να εμπλουτιστούν οι τοπικές κοινότητες με τη μεγαλύτερη συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων στη ζωή των κοινοτήτων. Η παρουσία των ανθρώπων αυτών είναι μια ευκαιρία. Αυτόν τον όρο τον έχουμε χρησιμοποιήσει πολλέ φορέ σε προηγούμενε συζητήσει. Μια ευκαιρία ανάπτυξη για όλου. Και για του ντόπιου και για του αλλοδαπού. Η συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών ε, οδηγεί σε αμοιβαίο σε πλούτο για όλου. Ε, η Εκκλησία ε, επιμένει στα εξή σημεία. Πρώτον, καλούνται τα κράτη να ευνοήσουν την ένταξη ως κοινωνική πρόοδο που ε, αποδέχεται και ε, προωθεί, προάγει την, ε, τον πολιτισμό του άλλου. Θα πρέπει δηλαδή τα στοιχεία των γλωσσικών γνώσεων και των οικονομικών επαρχόντων να μην είναι τα κριτήρια ένταξης των μεταναστών αυτών, αλλά να επιτρέπεται η οικογενειακή τους επανένωση και να επιτρέπεται η παραμονή του στην εθνική επικράτη εφόσον ήδη διαθέτουν μια μακρά παραμονή. Επίση, θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη απέναντι στου πρόσφυγε μετανάστε και του άσυλο μέσω τη χρηματοδότηση διαπολιτισμικών ανταλλαγών. Την ανταλλαγή καλών πρακτικών για το θέμα μεταναστών και προσφύγων. Διασφαλίζοντα ότι οι κρατικέ προκηρύξεις δημοσιεύονται και στι γλώσσε των μεταναστών και προσφύγων και προ όφελο των τοπικών κοινοτήτων. 20. Ενθαρρύνονται τα κράτη-μέλη να ε, προστατεύσουν τους αλλοδαπούς που έχουν αποδράσει από περιοχές με εχθροπραξίες πολέμους και πολεμικές συγκρούσεις. Να συμμετάσχουν λοιπόν σε προγράμματα για την ενίσχυση των χωρών προέλευσής τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με την ε, ε, κατασκευή δομών και υποδομών στις χώρες προέλευσης και την περαιτέρω εκπαίδευση των μεταναστών και προσφύγων κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό με τι συνθήκε που προσφέρονται και στου ίδιου του πολίτε μια χώρα και την ταχεία επανένταξή του στι χώρε προσελευσή του και την αγορά εργασία του. Με συγχωρείτε που ξέχασα να λέω το next σε κάθε επόμενη διαφάνεια, αλλά τέλο πάντων έλεγαν ε, προωθώ, ενισχύω και εργαζόμαστε μαζί. Ε, αυτό είναι το επόμενο. Ε, το σύνολο των 20 αυτών σημείων παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικές περιστάσεις. Το τελικό κείμενο σε διαφορετικές γλώσσες έχει υποβληθεί στο Προεδρείο τη Επιτροπής σας, στη Γραμματεία μάλλον της Επιτροπής σας, για να λάβετε γνώση. Ε, τελευταίο, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Και συγχωρείτε που σας πίεσα να τελειώσετε γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πάντως να αναφέρω κάποια πράγματα στους ε, συναδέλφους ε, γιατί και εγώ έκανα μια γρήγορη εισαγωγή. Να εξηγήσω ότι το τμήμα αυτό ε, για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες της Αγίας Έδρας από τον Πάπα όταν ακριβώς άρχισε να εντείνεται η κατάσταση και η Εκκλησία παρενεύει πολιτικά, αν μου επιτρέπετε, στο θέμα, αλλά συζητάμε με την γραμματεία και αν μου επιτρέπετε και ο πάτερ Χερνάντες, ο οποίος είναι εδώ ως νούντσιος του Βατικανού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα σημεία τα οποία είπατε έχουν κοινά σημεία με τα δικά μας δεν είναι ότι ξαφνικά ήρθατε εδώ πέρα ε, μία μέρα και ιδιαίτερα επίσης ε, βοηθάει τους πρόσφυγες ε, και τους μετανάστες σε πολλές χώρες. Αυτά θα ήθελα να αναφέρω και θα αναφέρω και κάποια άλλα πράγματα μετά. Να περάσουμε τώρα στους βουλευτές που θα ήθελαν ίσως να πούν δύο λόγια ή να κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Ξεκινάμε την κυρία Κιέγγε. Ευχαριστώ, Κλοντ. Όχι τόσο ερωτήσει θα ήθελα να κάνω με την παρέμβασή μου, αλλά να υπογραμμίσω τι ομοιότητε μεταξύ τη δουλειά που μα παρουσιάστηκε και σα ευχαριστώ εκ βαθέων για την πολιτική σα αυτή πρόταση. Και παρακολουθούμε με προσοχή τα όσα κάνετε, αλλά ήθελα να επιστρέψω λίγο έτσι γρήγορα ε, στο 2013 όπου όλα άρχισαν λίγο να αλλάζουν, χάρη στη δράση του Παπα Φραγκίσκου τον Ιούλιο του 2013, πήγε στη Λαμπεντούζα και για πρώτη φορά έριξε άνθη στα νερά της θάλασσας για να θυμηθούμε ότι οι μετανάστες είναι άνθρωποι και χάνουν στη θάλασσα τη ζωή τους. Προηγουμένω μιλάγαμε για αυτού του παράνομους μετανάστε, λες και ήταν φαντάσματα που στα θεσμικά μας όργανα δεν είχαν καν θέση. Όλα αυτά άρχισαν να αλλάζουν μετά τη δική του παρουσία στη Λαμπεντούζα και τη ρήψη ανθέων στη θάλασσα. Έτσι έγινε σαφής ο ρόλος του. Η εικόνα και η προσωπικότητά του έχει επηρεάσει και στις πολιτικές, πολιτικές μας επιλογές, κυρίως στην ε, έρευνα και διάσωση. Αυτό στην Ιταλία οδήγησε στην δημιουργία του προγράμματος Mare Nostrum. Το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό εγχείρημα με 150.000 ανθρώπους να διασώζονται και σε ένα ψήφισμά μα περιλαμβάνονταν πολλά σημεία που μοιάζουν με όσα μα είπατε. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Ευρωκοινοβούλιο για την ολιστική προσέγγιση τη διασώση στην Μεσόγειο. Πρέπει να πω ότι είμαι ευτυχή, διότι βλέπω σημεία στο κείμενό σα που όχι απλώς εκφράζουν τις βασικές ε, αξίες του καθολικισμού, αλλά και αξίες ε, που δείχνουν να σέβονται το διεθνές δίκαιο και γενικότερα για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι πραγματικά διορατικότατο το κείμενό σας και μοντέρνο, σύγχρονο. Είναι ανθρωπιστικές οι αξίες που εκφράζεται και τώρα κάποιες συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Τα τέσσερα σημεία που μας απαριθμίσατε. Το υποδοχή, προστασία, προώθηση και επανένταξη, όλα αυτά είναι εξαιρετική σημασίας. Η προοπτική της ασφάλειας θα πρέπει πάντοτε να προέχει της εθνικής ασφάλειας, όπως και τα αναλύωτα δικαιώματα των ε, μεταναστών το δικαίωμα στο άσυλο και στην προστασία έχετε συμπεριλάβει την διασπορά την... Που, δεν που δεν την καλύπτουν πολλές φορές τις ζητήσεις τους στα κάτι μέλη. Αυτή τη διασπορά την έχουμε συμπεριλάβει στα κείμενα του Ευρωκοινοβουλίου όταν συζητούσαμε και για το Σύμφωνο Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης και αναγνωρίζοντας το ρόλο της διασποράς αυτής. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτήν την διάβια και διορατικότητα. Το άλλο βασικό σημείο είναι ε, η ηθαγένεια αλίμονο. Είναι πολλά αυτά που ακόμη απομένουν να γίνουν και στη χώρα μου την Ιταλία και σε αλλα κρατημέλη. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα του πολίτη στα άτομα αυτά που δεν έχουν γεννηθεί στο έδαφο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω λέτε κι εσεί, πρέπει να συνεργαστούμε και ξέρω πόσο αφοσιωμένοι είστε σε αυτόν τον σκοπό για να προσφέρουμε το δικαίωμα του πολίτη, την ηθαγένεια. Ε, και κάτι ακόμη που θεωρώ διορατικότατο και το εκτιμώ αδιαιτέρω. Στο σημείο που ζητάτε ω Καθολική Εκκλησία, στο 17, να διασφαλίσετε πάντοτε η ανεξιθρησκεία και στο δόγμα και στην εξάσκηση των θρησκευτικών δικαιωμάτων για όσους ετούντε άσυλο πρόσφυγε ή μετανάστε φτάνουν σε μια χώρα ασχέτω με το καθεστώ του καθεστώ ω προ τη μετανάστευση. Δεν ζητάτε να ε, αλλαξοπιστήσουν και να γίνουν καθολικοί. Ζητάτε την ανεξιθρησκεία. Αυτό το θεωρώ εξαιρετικό για να περάσουμε σε αυτή τη φάση προ το διάλογο. Σα ευχαριστούμε λοιπόν και θα φροντίσουμε να αποφυσαυρίσουμε το κείμενο αυτό. Um, Ευχαριστώ, Σεσίλ. Κυρία Σπινέλη. Να ευχαριστήσω τον ε, πατέρα Μπάντζο και για το πρόγραμμα δράσης και θα πρέπει να ευχαριστήσω και τον Ποντίφικα που ήταν η πηγή έμπνευσης. Ιδίως ως προς κάποια σημεία ουσίας που στέκονται στις ανάγκες των μεταναστών και προσφύγων. Το γιους σόλι, το δίκαιο του εδάφους, η κοινωνική ένταξη, επανένωση των ε, ε, οικογενειών με διευρυμένη έννοια. Η ε, επανεξέταση των ασφαλών χωρών προέλευσης, τα δικαιώματα που θα πρέπει να προσφέρονται στους μετανάστες πρόσφυγες και άσυλο, ασχέτως του νομικού τους καθεστώτος. Είχα μερικές ερωτήσεις για μερικά συγκεκριμένα σημεία του κειμένου. Πρώτον, η πρόσκληση που απευθύνεται στις ε, επισκοπικές έδρες να αποστείλουν το πρόγραμμα αυτό στις οικίες κυβερνήσεις, ιδίως τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για τα θέματα αυτά. Τι να κάνουν οι επισκοπικές αυτές σύνοδοι κάποιων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκονται σε χώρες που είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές, για να το πω με έναν εφημισμό. Την Πολωνία και την Ουγγαρία, ας πούμε. Τι να κάνουν σε αυτές τις δύο χώρες οι σύνοδοι των επισκόπων. Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά την νομοθεσία, τον νόμο. Λέγεται στο κείμενο ότι η μετανάστευση πρέπει να είναι μια διαδικασία ε, τακτική και να βασίζεται στην νομοθεσία της κάθε εμπλεκόμενης χώρας. Αυτό που λίγο με ξαφνιάζει είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές μνήες στη διεθνή, στις διεθνείς συμβάσεις, στο διεθνές δίκαιο, με την εξαίρεση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Νηπίων. Δεν γίνεται αναφορά σε έναν νόμο, μια συμβάση που θεωρώ θεμελιώδου σημασία και εγώ προσωπικά. Δεν αφορά μόνο την διαφυγή από δικτατορικά καθεστώτα ή πολέμους, αλλά το δικαίωμα να εγκαταλείψει κανείς την οποιαδήποτε χώρα, ε, συμπεριλαμβανομένη της δικής του, όπως αναφέρεται στην οικονομική, οικουμενική διακήρυξη των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου, αυτό είναι, υπερέχει ακόμη και τον ε, του τι συμβαίνει σε περιπτώσεις πολέμου. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να εγκαταλείψει τη χώρα του. Και κάτι άλλο το τελευταίο. Στο σχέδιο που μας προτείνεται, όταν λέγεται, ε, όταν υπάρχει αυτή η μνήμα για την ε, προστασία, την αξία της προστασίας της προσωπικής ενός ατόμου, θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή αντιστοίχηση μεταξύ της ασφάλειας της προσωπικής, θα προσέθετα και της αξιοπρέπειας της προσωπικής και των μεριμνών για την ασφάλεια μιας χώρας. Αυτό είναι ένα πολύ λεπτό θέμα. Και εκεί, κατά την άποψή μου, πρέπει να γίνει μια αναφορά στο διεθνές δίκαιο, που είναι πολύ ακριβές ως προς τη σωστή εξισορρόπηση των δύο αυτών προτεραιοτήτων. και φροντίζει να μην δοθεί ε, μεγαλύτερο βάρος στις ε, μέρημνες ασφάλειες μιας χώρας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Μπάρμπαρα. Συνα... Συνάδελφε, ε, μετά την ε, δημόσια αυτή ακρόαση θα έχουμε μια συνέχισε και κλεισμένο το θηρόν της συνεδρίασης. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας θέλω παρακαλώ να είστε πολύ λακωνικοί. Δύο ακόμη ομιλήτριες θα λάβουν το λόγο, η κυρία Ιντβελτ και η κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Μα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Μπάτζο ε, δεν ε, υπενώ συχνά την Καθολική Εκκλησία όπως ξέρετε. Αυτή τη φορά εκτιμώ την προσπάθειά σας. Ημών και του Πάπα. Και πολλά από τα 20 σημεία είναι ταυτόσημα με τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις απόψεις του κόμματός μου και μου. Βλέπετε λοιπόν ότι οι αξίες δεν είναι μόνο πόλιο του χ ή του ψ, αλλά καμιά φορά είναι κοινέ, αν θέλετε. Τα στηρίζω λοιπόν όλα αυτά και ελπίζω οι κοινέ μας προσπάθειες να αποδώσουν. Όμως θεωρώ ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για να επιτύχουμε αυτά τα 20 σημεία είναι η πολιτική με όμικρον γιώτα και με ήττα. Και η πολιτική με όμικρον γιώτα που εμποδίζουν τα αποτελέσματα είναι η πολιτική που είναι και καθολική και χριστιανοδημοκράτες. Ε, κάποιοι από αυτούς ε, είναι, θα έλεγα, πώς να το πω, οι ε, σκληρότεροι αντίπαλοι μιας ανθρωπιστικής πολιτικής. Μιλάω για τους χριστιανοδημοκράτες Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία, τη Βαβαρία και αλλού. Και αναρωτιέμαι το τι ε, μπορείτε να κάνετε για να ασκήσετε την επιρροή σας σε αυτούς. Γιατί είναι προφανές ότι κυνηγούν την ακροδεξιά ψήφο και γύρουν ξενοφοβικά συναισθήματα για εκλογικά ωφέλη. Ε, τόσο νόμιζα ότι είχα δικαίωμα να έχω την άποψή μου. Τέλος, αυτό νομίζω ότι οδηγεί σε κάτι το οποίο μας δείχνει πώς έχει οδηγηθεί το κλίμα και επί χριστιανοδημοκρατικής κυβέρνησης. Το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στη Βιέννη την πρωτοχρονιά ε, ήταν ένα κοριτσάκι ονόματι Ασέλ από μουσουλμάνους γονείς και η γέννησή της ε, βεβαίως ε, έγινε δεκτή όχι μόνο από συγχαρητήρια αλλά από ρατσιστικό μίσος κατά ενός νεογέννητου κοριτσιού και βεβαίω εκτιμώ το ότι μίλησε εναντίον αυτού του γεγονότος ο Πάπας, αλλά πρέπει να υπενθυμίσει και σε κάποιους πολιτικούς, όχι μόνο τους χριστιανοδημοκράτες, ε, τις αξίες τους. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνος τρόπος ε, να επιτύχουμε τα 20 σημεία τα οποία στηρίζω πλήρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Birgit. Ευχαριστώ. Εγώ θα είμαι πιο λακωνική γιατί με κάλυψε η Σόφη στο τελευταίο της σχόλιο. Μερικές ε, καθολικές ε, χριστιανοδημοκρατικές ε, κυβέρνησης χώρες και περιοχές απορρίπτουν κάθε μορφή σε ελληνική. Έχουμε δύο παραδείγματα. Στην Ουγγαρία έχουμε 3,8 εγγεγραμμένους καθολικούς και στην Πολωνία οι νέες στους 10 πολίτες δηλώνουν καθολικοί. Επιπλέον, όχι μόνο δεν θέλουν πρόσφυγες οι χώρες αυτές, αλλά αποποιούνται κάθε ευθύνη ό,τι αφορά την, το σύστημα επανεγκατάστασης. Δεν ενεργοποιούνται ούτε στη μετεγκατάσταση ούτε στην ευεγκατάσταση. δεν έχουν στρατηγική ε, κοινωνικής ένταξης και μερικές ε, συνθήκες σε καταβλισμούς προσφύγων είναι άθλιες ε, και Μάλιστα θέλουν να γύρουν φράχτες και τείχους γιατί δεν θέλουν ούτε ένα πρόσφυγα στο έδαφος τους. Ερωτώ λοιπόν, πολύ ωραίο ότι έχουμε κοινή θέση και συμφωνούμε και κάθε φορά που συναντώ εκπροσώπους της Καθολικής Εκκλησίας διαπιστώνω ότι έχουμε κοινέ απόψεις ε, και σύμπνοια και χαίρομαι. Ερωτώ όμω, εσεί τι κάνετε και τι μπορείτε να κάνετε για να συμβάλλετε προκειμένου να αλλάξει η νοοτροπία σε αυτέ τι περιοχέ και χώρε. Τι μπορείτε να κάνετε σε συνεργασία με τι ε, κοινότητέ σα στι χώρε αυτέ. Υπάρχει κάτι που θέλετε και δύναστε να κάνετε προκειμένου να στηρίξετε αυτέ τι κοινότητε που υπάρχουν και σε χώρε όπω η Πολωνία που θέλουν ε, επιθυμούν να στηρίξουν και να εντάξουν κοινωνικά τους πρόσφυγες, αλλά δεν έχουν τους πόρους για να το υλοποιήσουν. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να κάνετε ή που κάνετε ήδη, απτά και συγκεκριμένα, ή διαβλέπετε κάποιες κοινέ προσπάθειές μας για να συμβάλλουμε στην υλοποίηση πρόοδου. Πολύ καλή ερώτηση, πολύ εύστοχη γιατί γνωρίζω και εγώ από ε, συνάντηση με τον, και συζήτηση με τον Πατήρ ε, Μπάτζο ότι υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα που θα, θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Παρακαλώ, δεσιμότητα να είστε λακωνικός στις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ε, θα απαντήσω στη γλώσσα που τέθηκαν και οι ερωτήσεις. Ευχαριστώ τους, την κυρία Κέγκε για την εκτίμηση που μας έδειξε και δεν έχω να πω τίποτα άλλο, το παρατηρήσει περισσότερο. Η κυρία Σπινέλη έθεσε κάποιε ερωτήσει. Συμφωνούμε ω προ την ανάγκη που έχει διαπιστωθεί ε, και σε ό,τι αφορά το, τον κατάλογο των ασφαλών χωρών. Αυτό θα πρέπει να αναθεωρηθεί με βάση τα κριτήρια επιλογής ε, για τη συμπερίληψη των χωρών στον κατάλογο. Ε, ε είπατε για την πρόσκληση που απευθύναμε στις επισκοπικές συνόδους με την επίδοση αυτού του εγγράφου του σχέδιου δράση των 20 ε, σημείων. Φυσικά οι κυβερνήσεις ε, είναι επιφορτισμένες με τις διαδικασίες ε, της διαπραγμάτευσης για το Παγκόσμιο Σύμφωνο και εμείς συμμετέχουμε με το έγγραφο αυτό στο διάλογο και θέλουμε να βοηθήσουμε τις επισκοπικές συνόδους αυτή τη διαδικασία γιατί μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα ήταν πολύ θετικά. Είχαμε περίπου 40 άμεσες συναντήσεις με εκπροσώπους επισκοπικών συνόδων και προσπαθήσαμε να προωθήσουμε τα σημεία του σχεδίου δράσης μας. Μάλιστα είχαμε πολύ άριθμες ε, συναντήσεις στις οποίες επισημαίνουμε ε, τα σημεία αυτά και σε ό,τι αφορά το Παγκόσμιο Σύμφωνο εμείς υποβάλαμε 20 προτάσεις με τα σημεία αυτά. Έχουμε ε, φυσικά κάποια σημεία για τα δικαιώματα των παιδιών, των υπείων και των παιδιών. Και μέσα στο έγγραφό μας θα βρείτε πολλές παραπομπές σε έγγραφα του ΟΗΕ, ε, της ε, Παγκόσμια Οργάνωση για την Εργασία, παρόλο που κάποια σημεία δεν αφορούν άμεσα τη μετανάστευση. Επίσης, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της μετανάστευσης, πολύ συχνά το εξηγώ στους φοιτητέ μου, ε, είναι ένα συμμετρικό δικαίωμα. Έχουμε το δικαίωμα να αποδημήσουμε από τη χώρα μας και να επιστρέψουμε, αλλά δεν έχουμε το δικαίωμα ε, ε, να εισέλθουμε μερικέ φορέ στο έδαφο μιας χώρας, οπότε αυτό το δικαίωμα είναι ασύμετρο. Θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό το δικαίωμα που έχει κανεί ε, για την αυτοεκπλήρωση και την οικογενειακή εκπλήρωση προσκρούει σε κάποια άλλα δικαιώματα και θα πρέπει να γνωρίζουμε με ποιου όρου θα πρέπει να ασκείται το κάθε δικαίωμα. Επίση αυτό που θα ήθελα να πω προσωπικά είναι ότι θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας θα πρέπει να ενεργούμε υπεύθυνα και να επιτρέπουμε σε όλους να επιτύχουν την αυτοεκπλήρωση. Και αν δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο, να δούμε πώς μπορούμε να δράσουμε, γιατί υπάρχουν κάποιες ασύμετρες καταστάσεις, κάποιες ασυμμετρίες. Γιατί σε μερικέ χώρε δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο, να υλοποιηθεί αυτή η αυτοεκπλήρωση. Σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλεια και εθνικής ασφάλειας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αρμονία που υπάρχει σε νομικό και διεθνές επίπεδο. Δεν μπορούμε να φέρνουμε σε αντιπαράθεση την προσωπική ασφάλεια με την εθνική ασφάλεια. Γιατί σε ένα κράτος έχουμε πολίτες και σε μια ανθρωπιστική φιλοσοφία στα δικιά μας το κράτος υπάρχει μόνο ως ένωση ανθρώπων, ως ένωση προσώπων το κράτος δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τα άτομα. Και αυτό που λέμε στο έγγραφο είναι ότι θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της προσωπικής και της εθνικής ασφάλειας. Και ο Άγιος Πατέρας στο μήνυμα της 14ης Ιανουαρίου που θα δημοσιευτεί την επόμενη Κυριακή τόνισε ότι η προσωπική ασφάλεια θα πρέπει να υπερέχει ε, της εθνικής. Για τις δύο αυτές ε, παρόμοιες ερωτήσεις ε, θα προσπαθήσω να τις απαντήσω. Θα έλεγα ότι αν μπορούμε να μιλήσουμε για ψηφοφόρους. Πρόκειται για πιστούς και ο καθένας έχει βεβαίως διαφορετικό ρόλο στην κοινωνία, άλλοι είναι εργαζόμενοι, άλλοι είναι πολιτικοί, άλλοι έχουν άλλο ρόλο. Και θα ήθελα να πω ότι χιλιάδες από αυτούς έχουν εμπλακεί άμεσα στην υποδοχή μεταναστών ε, και προσφύγων και στην ένταξή τους και πρέπει να πω ότι είναι προφανές στην Ευρώπη και αλλού ότι η εμπλοκή της Καθολικής Εκκλησίας είναι συνεπής εδώ και χρόνια και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε χιλιάδες εργαζομένους που υποδέχονται εκατομμύρια ανθρώπους και προσπαθούν να τους εντάξουν και επενδύουμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ και ευχαριστούμε για όλα αυτά χάρη στους ε, πολλούς ε, δόρητες ε, που εμπιστεύονται την Καθολική Εκκλησία. Και χαιρόμαστε για το ότι βρήκαμε καλούς εταίρους σε άλλες εκκλησίες, σε άλλες ομολογίες και σε άλλες θρησκείες που συνεργάζονται μαζί μας. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερος στο πλαίσιο του διαλόγου που ανέφερε η κυρία Κιέγγε, διαθρησκευτικού διαλόγου Ο καθένα βεβαίω ε, δικαιούται να έχει την άποψή του και ε, για να αλλάξει η άποψη πρέπει να δώσουμε και κάποιον λόγο. Και η καθολική πολιτική επίση Ο Πάπας ε, είναι ρητό, νομίζω, σαφής και φέτος και πέρσι μίλησε και φέτος θα το κάνει για τις αρχές μας και το τι ζητάμε από την καθολική κοινότητα και τους καθολικούς ηγέτες και τους πολιτικούς. Τώρα ξέρετε πως η διαδικασία της αλλαγής, ε, της νοοτροπίας και του να επιτύχουμε μια συνένεση και βεβαίως να θέσουμε τα πράγματα σε ένα πλαίσιο όπου έχουμε μια συγκεκριμένη κατάσταση και βέβαια να αντιμετωπίσουμε τον φόβο, τον πραγματικό φόβο των ανθρώπων. Ίσως ε, να μην είναι ε, ο λόγος ε, του φόβου πραγματικός, αλλά ο φόβος εξακολουθεί να είναι πολύ πραγματικός και εκεί πέρα ακριβώς πρέπει να εργαστούμε. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε σε όλες τις χώρες και θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όχι μόνο κάποιες, Ε, και θα έλεγα ότι πρέπει να τα θέσουμε αυτά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και να θέσουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και τον φόβο, όπως είπα, που είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε μαζί τώρα. Αυτό το οποίο είπα πριν για να αλλάξει το αφήγημα είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε από κοινού. Δεν μπορούμε κάθε μέρα να διαβάζουμε αρνητικές ειδήσει για μετανάστες πρόσφυγες κτλ. φαίνεται ότι αυξάνεται ε, το αρνητικό αφήγημα και δεν μας επιτρέπει να δούμε τις ευκαιρίες που πάντα υπάρχουν γιατί βεβαίω δεν αποκαλύπτονται εύκολα, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν, τις ανταλλαγές των πολιτισμών, την ε, δυνατότητα να αναπτυχθούμε έτσι από κοινού. Και βεβαίως είτε θα αναπτυχθούμε από κοινού είτε δεν θα αναπτυχθούμε καθόλου. Πρέπει να δούμε λοιπόν ε, μια ευρύτερη εικόνα. Και αυτό το οποίο είπε επίσης ε, και ο Πάπας, ε, απευθυνόμενος προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστια ευθύνη. ακριβώ γιατί εδώ πέρα έχουν βρει τον καταλληλότερο τόπο από τα ανθρώπινα δικαιώματα. και θεωρώ πως αυτό δεν είναι μόνο αποστολή της Καθολικής Εκκλησίας, είναι αποστολή της Ευρώπης. Γι' αυτό ακριβώς δεχτήκαμε την πρόσκλησή σας ε, να έρθουμε εδώ και από τώρα να ξεκινήσουμε να έχουμε στενότερες ε, σχέσεις. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για οποιαδήποτε άλλη πρόταση έχετε τα στοιχεία μου και ευχαρίστως θα σας δώσουμε και άλλα δεδομένα. Σας ευχαριστώ. Ξέρω τώρα πως ο χρόνος τελείωσε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ειλικρινιά σας. Τώρα... κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, το βάρος ε, τώρα δόθηκε στο Παγκόσμιο Σύμφωνο του ΟΗΕ και θα έχουμε τουλάχιστον δύο τέτοιες συνεδριάσεις μία τον Φεβρουάριο και μία με την Επιτροπή Υπερυπολογισμού και όπως μας υπενθύμησε εδώ και ο πατέρας Μπάτζο Καθολική Εκκλησία και άλλες εκκλησίες παρέχουν πολλές υπηρεσίες οπότε να γνωρίζουμε και τον μεγάλο πρακτικό ρόλο που παίζουν στα περισσότερα κράτη-μέλη δεν είναι μόνο πολιτικό το ζήτημα είναι και θέμα προϋπολογισμού και ένταξης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν, Πάτερ. Και και την συνεργασία μαζί σας στο μέλλον και να μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μας ε, στον Ποντίφικα. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα.